Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, μεγάλη μου χαρά σήμερα που είμαι εδώ. Ελπίζω να περάσετε καλά τις διακοπές. για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας μετά από μια ευχάριστη ε, περίοδο ανάπαυσης. Ελπίζω να μην πάθατε κι εσείς τίποτα όπως και εγώ ε, έπαθα στο βόλεϊ, παίζοντας βόλεϊ. Θα με δείτε με εκείνο το αμαξίδιο που είναι και πολύ γρήγορο. Πολύ το ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, ε, καλώς ορίσατε όλοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Στο σημείο 10 της ημερήσης διάταξης είμαστε. Κοινή βάση φορολογική η φορολογία εταιριών και κοινή ενοποιημένη βάση φορολογία εταιριών. Οι συγχυτές μα είναι ο κύριο Τάγκα και ο κύριο Λαμασούρ. Και σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο, τα σχέδια εκθέσεων και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Πολ Τάγκ και μετά στον Αλέν, αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτή τη σειρά. Πολ, έχεις πρώτος το λόγο 10 λεπτά maximum και οι δύο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Να πω ότι στην ημερήσια διάταξη έχουμε δύο χωριστά ε, σημεία στην ημερήσια διάταξη, το 10 και το 11. Ο Αλέν και εγώ όμως πιστεύουμε πως αυτά ε, τα δύο σημεία είναι αλληλένδετα και γι' αυτό αποφασίσαμε να τα εξετάσουμε ως τμήμα ενός, ενός πακέτου και να μπορέσουμε έτσι να τα συνδυάσουμε και να τα συγχρονίσουμε όσο γίνεται περισσότερο και έτσι να φτάσουμε και να ολοκληρώσουμε την εξέταση των δύο φακέλων ταυτόχρονα. Κοινή βάση εταιριών χωρίς ενοποίηση δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως ε, αν, είχαμε, αν έχουμε ενοποιήσει και γι' αυτό και γι' αυτό η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο προτείνουμε και οθούμε την ιδέα των τριών ψη ταυτόχρονα. Η πρόταση CCTB ε, ε, δεν είναι ένα συνοθήλευμα είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο. είναι τη μετακίνηση από μια ε, βάση πηγή σε μια ε, βάση προορισμό. Αυτό αποτελεί πλέον αναγκαιότητα γιατί τα συστήματα των, ε, της φορολογίας εταιριών έχουν ξεπεραστεί. Αν προσπαθούμε να βρούμε την τοποθεσία των κέντρων κερδοφορίας είναι πολύ δύσκολο να το γιατί γιατί ακριβώς οι δομές έχουν γίνει αόριστες όσον αφορά την οικονομική, ε, το οικονομικό οικοδόμημα. Ε, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ποια είναι η πραγματική, η φυσική τοποθεσία της ε, κάθε εταιρεία. Ο καιρός αυτός έχει περάσει προπολού και γι' αυτό και χρειάζεται μια κοινή βάση φορολογίας των εταιριών και η CCTB αυτό υπόσχεται ακριβώς. Και πάλι ε, είναι απαραίτητο, ας πούμε, στη χώρα μου, στην Ολλανδία, έχουμε γίνει μια χώρα διέλευση για τις ε, χρηματοπιστωτικές ροές δηλαδή ε, κεφάλαια, μερίσματα, ε, επιτόκια, αλλά και η απόδοση από την πνευματική ιδιοκτησία και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά περνάνε από την Ολλανδία, πράγμα που δείχνει με ξεκάθαρα το πρόβλημα με τα σημερινά συστήματα φορολογίας εταιριών. Η CCTB λοιπόν απαντά σε αυτό το πρόβλημα γιατί δεν επιμένει στην αρχή της πηγής αλλά στην αρχή του προορισμού αντιμετωπίζοντας έτσι το πρόβλημα. και γι' αυτό και το σύστημα αυτό προορισμού των κερδών είναι ένας σωστός τρόπος για να μπορέσουμε τη φορολογία εταιριών να τη φέρουμε πλέον στον 21ο αιώνα. Επίσης έχουμε πολιτικό πρόβλημα. Ε, εδώ παίρνω τη δική μου χώρα ως παράδειγμα, αλλά υπάρχουν μικρότερες χώρες που παίζουν ε, το ρόλο της διάβρωσης της φορολογικής βάσης. Παίζουν αυτό το παιχνίδι του ε, προσπάθειας προσέλκυσης ροών προς την ε, λόγω χώρα. Για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία μαζί έχουν ε, περισσότερες άμεσες ε, ξένες επενδύσεις από ότι η ΙΠΑ και η Ιρλανδία περισσότερο από τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Και αυτό βέβαια βασίζεται στις, στα διάφορα οικοδομήματα. Η CCTB λοιπόν αντιμετωπίζει αυτό το είδους το πρόβλημα. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση για την Ευρώπη για εξυγχρονισμό του συστήματος φορολογίας εταιριών ώστε να μπούμε στον 21ο αιώνα, να σταματήσουν αυτού του είδους τα ε, οικοδομήματα αλλά και να φτιάξουμε έτσι ένα ισότιμο πεδίο γιατί οι ευκαιρίες για φορολογικό σχεδιασμό είναι περισσότερες για τις μεγάλες εταιρείες από ό,τι για τις μικρές. Είδα διάφορες μελέτες για διάφορες χώρες που δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν ένα τρίτο περισσότερο ε, φόρους από ό,τι οι μεγάλες εταιρείες. Εάν δεν σας πείθει το ότι είναι άδικο, θα πρέπει να, σίγουρα να πούμε ότι αυτό δεν είναι επαρκές. Δεν είναι ένα ισότιμο πεδίο για τις εταιρείες μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις πολυεθνικές, τους ομίλους. Γι' αυτό και καλό το ΕΛΚΑ μαζί με τον Αλέν Λαμασούρ να καλωσορίσει αυτό, αυτή τη μεταρρύθμιση. Τούτου λεχθέντος υπάρχει μια μεγάλη παράληψη που έχει ε, εξεταστεί από τον ΩΣΑ. Μάλιστα, το πρώτο σημείο δράσης στον ΠΕΠΣ ήταν η πρόκληση της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. Είναι το πρώτο σημείο δράσης δεν ήταν ένα σημείο δράση όντω, γιατί ο ΣΑ ανέβαλε τη συζήτηση, συν, ε, συγκάλεσε μια task force και το έβαλε στο ράφι για άλλα πέντε χρόνια. Εμείς όμως γιατί περιμένουμε άλλα πέντε χρόνια, όταν γνωρίζουμε ότι η Google, το Facebook, η Amazon είναι παρόντες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όλοι χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους και ταυτόχρονα επειδή δεν εντάσσονται στο φορολογικό σύστημα αποφεύγουν τη φορολογία. Τόσο ο Αλέν Λαμασούρ λοιπόν όσο και εγώ πιέζουμε εδώ ώστε να ενταχθεί στην ε, έκθεση αυτή η ιδέα της φορολόγησης των ψηφιακών ε, πλατφορμών. πρώτα στην έκθεση CCTB, την κοινή βάση φορολογίας εταιριών, έχουμε ορίσει την ψηφιακή παρουσία ώστε οι ψηφιακές πλατφόρμες που είναι παρούσες εδώ να οφείλουν να καταβάλουν τους φόρους τους στις χώρες όπου χρησιμοποιούνται. Ας πούμε η Google χρησιμοποιείται στη Γερμανία, άρα θα πρέπει να πληρώνει φόρους στη Γερμανία και μετά έχουμε και μια διαφορετική φόρμουλα με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα μας απασχολήσει βλέπουμε μια πρωτοβουλία και από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Δεν μπορεί να περιμένουμε ακόμα πέντε χρόνια όπως προτείνει ο ΑΣΑ. Δεν χρειαζόμαστε task force, πρέπει να συζητήσουμε ιδέες για το πώς θα το κάνουμε αυτό και πώς θα συμπεριληφθούν οι ψηφιακές πλατφόρμες στο σύστημα φορολογίας εταιριών. Αυτή είναι λοιπόν μια παράληψη που πρέπει να διορθωθεί μέσα σε αυτή την πρόταση και έπειτα ε, το CCTB είναι ένα στεναρό και σύγχρονο σύστημα φορολογίας εταιριών. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο είναι στεναρό, αλλά είναι και απλό. Αν δούμε άλλα συστήματα φορολογίας εταιριών όπως στη χώρα μου και έχω ασχοληθεί με αυτό στο Εθνικό Κοινοβούλιο, ε, όλο και περιπλέκεται γιατί κάθε χρόνο προστίθεται μια εξαίρεση ένας κανόνας και πάντα αυξάνεται, μεγαλώνει, ποτέ δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται. Και αυτό είναι το καλό αυτή τη πρόταση. Πρόκειται για μια φορολογική μεταρρύθμιση που είναι απλοποίηση. Είναι απλό λοιπόν και ε, ε, στεναρό το σύστημα αυτό που προτείνουμε και γι' αυτό το λόγο στην έκθεση προτείνουμε ένα χαμηλότερο κατόφλι, δηλαδή 40 εκατομμυρία και αργότερα προτείνουμε να καταργηθεί. Και ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να ε, ωφελούνται μόνο οι μεγάλες εταιρείες από ένα απλό, απλούστερο σύστημα φορολογίας. Να χαμηλώσουμε το κατόφλι και αργότερα να το καταργήσουμε, αν είναι καλό όντως το σύστημα. Και πιστεύουμε πως είναι να μην αφήσουμε να ωφεληθούν μόνο οι μεγάλες εταιρείες και κυρίως όταν σκεφτούμε ότι ορισμένες από τις μικρότερες εταιρείες ε, θα ε, μεγεθυνθούν, θα επεκταθούν, θα εξάγουν. Αυτές οι εταιρείες θα έχουν μεγάλα ωφέλη εάν ενταχθούν σε ένα κοινό, κοινή βάση φορολογίας εταιρεών. Μια τελευταία παρατήρηση, αυτό που βλέπουμε Έχουμε ανταγωνισμό φορολογίας αυτή τη στιγμή, γιατί οι χώρες ε, ασκούν διάφορες πολιτικές, άσχετα με το ποιες θα είναι οι επιπτώσει για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να περιοριστεί και γι' αυτό προτείνω στην εκθεσή μου ένα μίνιμουμ ε, βάρο, φορολογικό βάρος του 8%. Αυτά είναι τα κύρια σημεία τη συζήτηση. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις και σχόλια με χαρά θα τα ακούσω και προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση ο Αλέν Λαμασούρ και εγώ όχι μόνο συνομιλούμε μαζί σας, αλλά έχουμε συνομιλήσει και με άλλα εθνικά κοινοβούλια. Πήγαμε στην Εστονία, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο και θα συνεχίσουμε το γύρο μας, περνώντας από τη Χάγη, το Παρίσι, τη Βερολίνο, το Βερολίνο και τη Σόφια. Γιατί πιστεύουμε πως είναι μια αξιόλογη πρόταση και με χαρά την προωθούμε. Ταυτόχρονα ξέρουμε πως υπάρχουν ανησυχίες και τις λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό και έχουμε αρχίσει αυτόν τον γύρο των χωρών και γι' αυτό και γίνεται η σημερινή συζήτηση να δούμε πώς η πρότασή μας θα μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητής για τη CCCTB, ο κύριος Λαμασούρ. Ευχαριστώ, αγαπητοί Πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω, όπως είπε και ο Παουλ Τάνγκ, ότι συνεργαζόμεθα στενά. Σαν να είμαι θα συνεισηγητέ για το συνολικότερο θέμα και με πολύ καλό και θετικό πνεύμα. Σε κάποια θέματα έχουμε βεβαίω πολιτικέ ε, διαφοροποιήσει και θα τι εξηγήσουμε φυσικά και η Επιτροπή θα αποφασίσει. Αλλά συμμεριζόμεθα την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτές τις δύο οδηγίες και συμφωνούμε ότι πρέπει να προσθεθούν και δύο πολιτικοί στόχοι στους στόχους της Επιτροπής. Η Επιτροπή παρουσίασε αυτά τα δύο κείμενα ως συμπλήρωμα και κατάληξη μιας σειράς πρωτοβουλειών που έχουν ήδη αναλυφθεί και ολοκληρωθεί εδώ και πάνω από δύο χρόνια ούτως ώστε να αποφευθεί ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός εντός της Ένωσης. Αυτό ήταν ο αρχικό στόχο. Αλλά εμεί θέλουμε να προσθέσουμε δύο ακόμη. Πρώτα απ' όλα να ωφεληθούν όλε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, πρώτα απ' όλα πιο μεγάλε, από ένα σύστημα φορολόγηση των κερδών που να είναι ενιαίο για την ενιαία αγορά, που να είναι σαφέ, που να είναι απλό, που να είναι δίκαιο και προσαρμοσμένο στην κατάσταση τη σύγχρονη οικονομία, που να είναι ένα πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και ο άλλο στόχο που προτείνουμε να προσθεθεί όπως σωστά είπε ο Πάουλ είναι να βρούμε τρόπο φορολόγησης της ψηφιακή οικονομίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και που σήμερα εποφελούνται από το γεγονός ότι επειδή δεν έχουν μόνιμη έδρα, permanent establishment σε μια χώρα της Ένωσης, καταφέρνουν να αποφύγουν να φορολογηθεί το μεγαλύτερο τμήμα των κερδών που ε, επιτυγχάνουν ιδίως ε, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπαθούμε λοιπόν να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και διαπιστώνουμε ότι μετά από μία περίοδο αδράνειας γίνεται ένας από τους κύριους στόχους η πρόθεση αυτών των δύο οδηγιών πολλών ε, εμπλεκομένων. Για παράδειγμα, η Εσθονική Προεδρία θέλει να το θέσει στην ημερήσια διάταξή τη, όπω ακούσαμε στο Τάλιν όταν πήγαμε. Και όπω είπε και ο νέο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία επίση, ο οποίο ανήγγειλε σε συμφωνία με τη Γερμανίδα ομόλογό του. Ακούσαμε λοιπόν ότι οι δύο χώρες μπορεί να υποβάλουν προτάσεις στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ για την ε, φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Έχουμε λοιπόν και τη δική τους τη βοήθεια για να προωθηθεί αυτό το θέμα που αντιμετωπίζει τόσες πολιτικές δυσχέρειες. Οι δύο οδηγίες, όπως είπε ο Πάουλ, είναι απόλυτα συνδεδεμένες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, συμφωνούν. Είναι σαφές ε, και από εμάς και για μας να εγκριθεί η πρώτη και όχι η δεύτερη οδηγία θα και την κατάσταση χωρίς να αποφέρει τα πλεονεκτήματα που αναμένουμε από αυτήν τη μεταρρύθμιση. Σημερίζομαι λοιπόν με τον Πολτάν ε, πολλές κοινέ απόψεις εκτός από δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα το θέμα του κατοφλίου. Οι σοσιαλιστές αρχικά και το ΕΛΚ αρχικά είχαν εντελώς διαφορετικές αφετηρίες θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό 750 εκατομμύρια ή αρκετά χαμηλά 40 εκατομμύρια μιλάμε πάντα για το, για το κύκλο εργασιών εγώ θα ήθελα να θέσω μια κάποια άλλη διάσταση γιατί θα πρέπει να υπάρχει κατόφλι διότι η μεταρρύθμιση αυτή θα βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις και γιατί να αστερίσουμε τα ωφέλη από τις μικρές επιχειρήσεις ή αυτή η μεταρρύθμιση θα περιπλέξει την κατάσταση, θα είναι επιπλέον μειονέκτημα. Γιατί τότε να θίξουμε τις πολυεθνικέ μας. Στη θέση της Επιτροπής βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα των μικρομεσαίων να ενταχθούν στο σύστημα. Αλλά οι επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν δεν έχουν την αναγκαία πείρα και θα ήταν πάντα δύσκολο. Και πρέπει να σκεφτούμε επίση και τι φορολογικέ αρχέ. Θα ήταν πολύ απλό να υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς και όχι δύο διαφορετικά. Και το άλλο θέμα, επί του οποίου τα κόμματά μας παραδοσιακά αποκλίνουν, είναι εφόσον αφορά τη φορολογική βάση. Το, γιατί να αφορά μόνο τη φορολογική βάση η πρότασή μας, γιατί να προτείνουμε και συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές μπορούμε να απορρίψουμε το καθορισμό οποιασδήποτε, οποιοδήποτε φορολογικού συντελεστή. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, να υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι, να πούμε ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να πληρώνουν τουλάχιστον τόσο και, μετά υπάρχει και μία τεχνική προσέγγιση. Η εναρμόνιση δεν έχει έννοια παρά μόνο εάν υπάρχει ένα ελάχιστο, ένας ελάχιστος φόρος που ε, καταβάλλεται. Τώρα τι σημαίνει ελάχιστος φόρος που καταβάλλεται ε, βεβαίως ε, είναι θέμα συζήτηση γιατί αν μια χώρα πει ναι βεβαίως έχω ελάχιστο συντελεστή μισό ή ενάμιση στην ουσία θα ήταν ε, εξαίρεση από το σύστημα όπως διαπιστώσαμε στο LuxLeaks. Τώρα κάποιες διευκρινήσεις για τις κυριότερες τροπολογίες που προτείνω να υπάρξουν στην οδηγία για το CCCTB Προτείνω, όπως είπε και ο Πολ στην οδηγία τη δική του, να υπάρχει μια τροπολογία που να προβλέπει την θέση σε ισχύ ταυτοχρόνως των δύο οδηγιών και αν δεν συμφωνήσουν 27 χώρες να εκινήσει ε, όσο ταχύτερα γίνεται μια διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας. Κάποια εθνικά κοινοβούλια είχαν κάποιες αντιρρήσεις συγκεκριμένα η αλλαγή φορολογικής βάσης θα γίνει εις βάρος των φορολογικών εσόδων κάποιων χωρών και εις όφελος κάποιων άλλων. Αν οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα δραστικές και κανείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε τέτοια στοιχεία, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να το κάνει. Προτείνω να δημιουργηθεί ένα ταμείο αντιστάθμιση που την πρώτη χρονιά θα χρηματοδοτηθεί από, την, ε, από τα επιπλέον ποσά που θα προέκυπταν για κάποια κράτη από το νέο σύστημα για να αντισταθμίσει ακριβώς ε, τη μείωση των φορολογικών εσόδων κάποιων άλλων κρατών. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε φάση εκπόνησης ενός προσωρινά βέβαια, προσωρινού βέβαια τέτοιου συστήματος για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές συντελεστών που θα προκληθούν από το σύστημα αυτό σε κάποια κράτη-μέλη. Όπως είπε ο Πολ επίσης, αν θέλουμε η φορολόγηση των κερδών να περιλάβει καλύτερα και τις ε, ψηφιακές συναλλαγές, θα πρέπει για να δούμε πώς θα κατανέμεται η φορολόγηση να μην πάρουμε μόνο τα, λεγόμενα, τα κριτήρια της Μασαχουσέτης, τα τρία του ΟΣΑ, αλλά να προσθέσουμε και ένα τέταρτο. Να είναι το επίπεδο των ε, δεδομένων ε, προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται από τους χρήστες και από τις πλατφόρμες. Και προτείνω μια μαθηματική φόρμουλα, που είναι μια πολύ δύσκολη βέβαια μαθηματική φόρμουλα. Εύκολα μπορεί να την επικρίνει όποιος να είναι, και από πλευράς μαθηματικής και από πλευράς πολιτικής. Αλλά θα ήθελα να εισαχθεί για να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Και όπως είπε ο Πολ, ο ΩΣΑ δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, πρέπει να τους υποχρεώσουμε να ξεκινήσουν την εξέταση του θέματος αυτού. Είναι λοιπόν μια φόρμουλα που κατά το ίμιση θα λάμβανε υπόψη τα στοιχεία που συλλέγονται και κατά το ίμιση τα στοιχεία που αξιοποιούνται. Επίσης, προτείνω κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο να κάνει μία αξιολόγηση της λειτουργίας αυτού του νέου καθεστώτος, λαμβάνοντας υπόψη και τις αξιολογήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και επίσης, μετά μια πενταετία, με βάση και τα πορίσματα που θα εξαχθούν από την εξέταση της πρώτης, της πρώτης περίοδου εφαρμογής, η Κομισιόν να κάνει νέες προτάσεις για την χρήση ενός τμήματος ή και όλου του ποσού που θα συλλεχθεί λόγω της κοινή αυτής φορολογικής βάσης να αποδοθεί λοιπόν ένα τμήμα ή το σύνολο αυτών των επιπλέον εσόδων στον ενωσιακό προπολογισμό. Είναι μια πρόταση, το συζητάμε Δηλαδή συζητάμε το θέμα των νέων ιδίων πόρων και του προπολογισμού της Ένωσης και την ίδια δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Συζητάμε λοιπόν τον ΦΠΑ τώρα που εδώ και 40 χρόνια έχει ενοποιημένη βάση θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εφόσον ήδη χρηματοδοτεί τον ε, προπολογισμό της Ένωσης. Εφόσον λοιπόν ε, ενοποιηθεί και η βάση φορολόγησης των εταιριών, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να αποδοθεί ένα τμήμα αυτών των πόρων στον προπολογισμό ή καλύτερα στη χρηματοδότηση της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Αλέλα Μασούρλη, ο Πρόεδρος. Τώρα οι σκιώδεις. Οκτώ λεπτά ο καθένας παρακαλώ. εκτός αν θέλουν ε, όπως οι άλλοι, να χωρίσουν το χρόνο μεταξύ περισσότερων μελών. Ο πρώτος είναι ο, ο κύριος Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές ε, για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει. Εκ μέρους του ΕΛΚ ε, ε είμαι σκιώδης στην εκθέση του Παουλ Τάγκ. Θα πρέπει, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να ασχοληθούμε και με το θέμα των εσόδων ε, των φορολογικών. Είναι το θεωρητικό πλαίσιο ε, και δεν ε, θα συνεισφέρει απαραίτητα στην αποδοχή από τα κράτη-μέλη. Οι παλιές προτάσεις του 2011 οδήγησαν σε μια σειρά συζητήσεων Ειδικά τις τελευταίους μήνες, μήνες είχαμε συζητήσεις με τις φορολογικές αρχές, τα κράτη-μέλη και οι επιπτώσεις ε, από τον ε, φόρο των εταιριών, για παράδειγμα, ε, έδειξαν ότι είχαμε πολύ σημαντική μείωση στα έσοδα των εσόδων. Υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, επειδή υπήρξε μια διαφορετική κατανομή λόγω αυτής της πρότασης, ε, υπήρχε αυτή η, ε, ο συμψηφισμός των πέντε ετών. Υπήρχαν ε, πολύ μεγάλες πιθανότητες εκπτώσεων λόγω της αναπτυξιακής πολιτικής που οδηγεί στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Επίσης, η πρόταση για την εφαρμογή βασίστηκε στην πρόταση της Κομισιόν. Έτσι ζητάω ο εισηγητής να πάει στα 40 εκατομμύρια ευρώ το όριο ε, του κύκλου εργασιών ε, και όταν θα έχουμε ένα ενιαίο φόρο εταιρεών στα κράτη-μέλη να αλλάξει πάλι σημαντικά ε, τα έσοδα των κρατών μελών. Ένας ενιαίος όμως φόρος εταιριών ε, όταν θα προκύψει ε, το να προκύψει ένας ενιαίος φόρος μάλλον εταιριών δεν είναι κάτι που αποδέχονται όλα τα κράτη-μέλη απαραίτητα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το πλαίσιο και να έχουμε και αρκετό χρόνο για να δούμε ποιες αλλαγές θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ε, πώς ε, θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Βέβαια, μακροπρόθεσμα έχει νόημα να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις εταιρείε, το οποίο ε, θα, είναι, θα έχει μια διάρκεια, να μην έχουμε δύο παράλληλα συστήματα εταιρική φορολόγησης, ας πούμε για μια εταιρεία η οποία είναι σε ισχύ, να έχουμε το εθνικό και το ευρωπαϊκό σύστημα ταυτόχρονα. Επίσης είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε από τώρα τις επιπτώσεις. Έχει γίνει κάποια εκτίμηση από την πλευρά της Κομισιόν. Όμως ε, δεν μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες ε, επαρκείς ε, για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν αλλάξουν τα πράγματα τόσο γρήγορα και τόσο εκτεταμένα, θα πρέπει να σκεφτούμε μια μακρά περίοδο προσαρμογής. Είναι επίσης ε, σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ε, η δυνατότητα κρατήσεων από την, ε, και εκτός λόγω της ανάπτυξης είναι κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα από τη φορολογία. Επίσης πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο οι ενισχύσεις που δίνονται κατά αυτόν τον τρόπο πολλές φορές γίνονται αντικείμενο κατάχρησης ή έχουν ε, περιορισμένες επιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το διερευνήσουμε γιατί δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Επίσης, οι εταιρείε που δεν έχουν τελικά κέρδη ε, ίσως δεν έχουν επιπτώσεις σε χρήμα, αλλά μπορεί να έχουν καλύτερη ανταγωνιστικότητα ή να μπορούν να επενδύσουν. Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Η πρόταση του εισηγητή να περιοριστούν οι εκτόσεις για λόγους έρευνας είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε. Όσον αφορά την απαλλαγή για την ε, καινοτομία και την ανάπτυξη, να πω ότι υπάρχει αυτό το μειονέκτημα που έχει να κάνει με τα ίδια κεφάλαια και τα ξένα κεφάλαια. Αυτό πρέπει να το ε, καταργήσουμε αν θέλουμε να πάμε παραπέρα. Επίσης υπάρχουν ε, νέοι ε, μηχανισμοί που είναι απαραίτητοι, οι οποίοι όμως είναι περίπλοκοι και μπορεί να έχουν ε, και αποτελέσματα ε, ανεπιθύμητα ή να δρουν και βάση του κύκλου της οικονομίας προκυκλικά. Δεν θα πρέπει λοιπόν φορολογικά να υπάρχει μειονέκτημα προς τα ίδια κεφάλαια. Αυτό θα πρέπει να το καταργήσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, να μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, περισσότερη από ότι με ξένα κεφάλαια, χωρίς να έχουμε μειωμένα φορολογικά έσοδα. Όσον αφορά στα ψηφιακά ζητήματα, έχει ε, ο εισηγητής ασχοληθεί πολύ με αυτή τη διάσταση. Έχουμε τις ψηφιακές ε, έδρες επιχειρηματικές έδρες. Ε, υπάρχει ένα πλαίσιο στη διαδικασία αυτής της ενοποίησης. Είναι σημαντικό λοιπόν ο νέος ε, εταιρικός φόρος των εταιριών να προσανατολίζεται προς την ψηφιακή εποχή. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στο σύστημα αλγορίθμους ε, και άλλα τέτοια ποσοστά και κλάσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στο σωστό φόρο. Επίσης, ο εισηγητής προτείνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ ως όριο για τα ψηφιακά συμβόλαια και τον όγκο περιεχομένου που έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες ε, και δημιουργούν τέτοια κέρδη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να μετρήσει αυτά τα νούμερα και υπάρχει ενδεχομένως ε, ανάγκη για ε, πράξη κατεξουσιοδότηση από την ε, Κομισιόν για αυτό το θέμα. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι ο εισηγητής ζητά από την Κομισιόν να προτείνει έναν ελάχιστο ενιαίο κοινό φόρο κοινή βάση φορολογίας εταιριών ε, υπάρχει το θέμα του Παναμά εδώ. Θέλουμε να δούμε αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό ε, καλό θα είναι να σκεφτούμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε, να μην είναι μόνο του στα κράτη-μέλη σε αυτό όσον αφορά στους φόρους, τον ΦΠΑ ε, και σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί όταν θέλουμε να στείλουμε κάτι στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για όλες τις ιδέες που έχετε καταθέσει στο τραπέζι και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτές. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω με μία παρέμβαση του σκιώδου ε, εισηγητού για την έκθεση του κυρίου Λασαμούρ και επέτα θα σας, θα σας ε, παραθέσω την ε, παρέμβαση της κυρίας Περβάνος Μπερές που η οποία ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα. Όπως ξέρετε, όπως μάλλον είχαμε επαφή με τις βελγικές αρχές μας αποκάλυψαν ότι 221 δις ευρώ έφυγαν για διάφορους φορολογικούς παραδείσους στο περασμένο χρόνο. Πάνω από το μισό του ΑΕΠ του Βελγίου. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό κοντεύει να φτάσει το σύνολο των αποταμιεύσεων των ε, ε, Βέλγων. Όπως και οι βελγικές εταιρείες έχουν πολύ λίγες, ίσως και καθόλου σχέσεις με το Μονακό και τα νήσους Καϊμάνα. και αυτό το παράδειγμα σας το δίνω, γιατί βλέπουμε έτσι πως ε, αυτές οι, αυτά τα εμβάσματα έχουν μόνο ένα στόχο να αποφύγουν την φορολογία και πιστεύω πως είναι πλέον ε, η κατάλληλη στιγμή να ξαναδούμε το σύνολο του συστήματος του φορολογικού. Πρόκειται για αστρονομικά ποσά που χάνουν κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη της Ένωσης και θα μπορούσαν αυτά να χρησιμοποιηθούν στην πραγματική οικονομία για να βοηθηθούν οι πολίτες ή για την κατασκευή υποδομών, νοσοκομεία, δρόμοι, σχολεία και ούτω καθεξής. Και μάλιστα συμφωνώ με τον συνάδελφο Λαμασούρ ότι κομμάτι αυτών των πόρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ήδη για να χρηματοδοτηθεί η Ένωση, είτε με σχέδια επενδυτικά, είτε με προγράμματα όπως το Horizon 2000 ε, ε, μάλλον στον ορίζοντα του 2020. Ε, αυτό το θέμα είναι υποσυζήτηση εδώ και καιρό. Το 2011 άρχισε η Ευρώπη να ασχολείται με μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών με στόχο να μπορέσουν οι εθνικές αρχές να ενοποιήσουν τα αποτελέσματά τους και να μπορούν αυτά να φορολογηθούν ανά κλάδο. Η Κομισιόν ξαναέθεσε αυτό το θέμα λοιπόν στη μερική Χαιρόμαστε γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές τον κύριο Τάγκο και τον Λαμασούρ που, είναι Έφτιαξαν πολύ ε, επικοδομητικέ εκθέσεις. Να επιμείνω, ας πούμε, εκεί όπου ο Πολ ε, ενίσχυσε κάποια στοιχεία στο κείμενο, όπως, ας πούμε, την ε, φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, γιατί ξέρουμε πως στο μέλλον αυτό θα γίνει και πρέπει εμείς να μπορούμε να συνοδεύσουμε αυτή τη μετατροπή, τη μεταμόρφωση της οικονομίας μας, έπειτα εναρμόνιση των ευρωπαϊκών ε, κανόνων φορολόγησης, ώστε να έχουμε μια ελάχιστη ευρωπαϊκή φορολόγηση φιλόδοξη για να αποφύγουμε τον προς τα κάτω ανταγωνισμό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό όλες οι εταιρείε να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες και όχι μόνο αυτές που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ συμφωνώ με τον κύριο Τάγκ, το σύστημα που θέλουμε να φτιάξουμε είτε θα είναι βιώσιμο και θα ισχύει για όλες τις εταιρείε είτε όχι. Το να βάζουμε έτσι ένα ψηλό ποσό, 750 εκατομμύρια ευρώ ως όριο, νομίζω πως δεν είναι λογικό. Αυτή η οδηγία είναι μια ευκαιρία για να φτιάξουμε μια νέα αγορά πιο ε, δίκαιη απέναντι στις ευρωπαϊκές εταιρείε, αλλά είναι και η ευκαιρία για να μειωθεί ο φορολογικός ανταγωνισμός που ζούμε καθημερινά ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να εξηγενθούν η δημόσια οικονομία αλλά και οι δυνατότητε επενδύσεων των κρατών μελών. με όλοι για πολιτική, είτε είμαστε αριστεροί είτε δεξιοί. Είμαστε πεπισμένοι πω το σύστημα δεν λειτουργεί πλέον και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να βρούμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Και οι δύο εκθέσεις που έχουμε επιτάπητος είναι ήδη πολύ θετικές. Και τώρα θα σας διαβάσω την ε, παρέμβαση της συντονίστριάς μας, της κυρίας Μπερβάνου Σεμπερές, που, όπως σας είπα ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα και θέλει να χαιρετήσει την εξαιρετική εργασία των δύο εισηγητών που είναι για εκείνη μια πολύ καλή βάση αφετηρίας. Ε, θέλουμε να Θέλει να υπογραμμίσει τέσσερα σημεία. Καταρχάς ε, την προσέγγιση σε δύο φάσεις που προτείνει η Κομισιόν. Φανταζόμαστε ποια είναι η λόγη που την όδησε να κάνει μια τέτοια πρόταση. Α, συγγνώμη. Α, ωστόσο, δεν θα πρέπει αυτή την πρόταση να τη στηρίξουμε, γιατί θα πρέπει μια κοινή βάση χωρίς ενοποίηση μπορεί αυτό να θέσει σε αφισβήτηση όλο το project. Δεύτερον, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την ψηφιακή οικονομία, να εξυγχρονίσουμε την ε, φορολογική ε, βάση, όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κεφάλαια των μεγάλων ε, γιγάντων του ίντερνετ, του διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να διορθώσουμε τις δυνατότητες που ανοίγονται ε, ε, να, μην να αποφύγουμε μάλλον τον κίνδυνο νέων ε, προβλημάτων μέσω αυτών των φορολογιών και έπειτα για τα κατόφλια υπάρχουν σημεία που πρέπει να προχωρήσουμε και η κυρία Μπερές ε, κατανοεί τα επιχειρήματα των ΜΕ και των ΔΕ, όμως είναι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μείνει αξιόπιστη και αποτελεσματική να αποφασίσει, είμαστε όλοι αιρετοί, πρέπει να δώσουμε, να λογοδοτούμε και η μηδενική φορολογία ή η φορολογία 12% θα ε, είναι μόνο, έχει το μόνο στόχο να αποφύγει, μάλλον να ελκύσει ε, κεφάλαια. Δεν θα πρέπει να φτιάξουμε έναν ε, μηχανισμό ελαστικό ώστε να πάψει αυτό ε, ο ανταγωνισμός ε, ο φορολογικός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η πρόταση του 2011 απέτυχε στο Συμβούλιο γιατί 28 χώρες δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν και να φτάσουν στην ομοφωνία που χρειαζόταν για τα φορολογικά θέματα και η επικαιρότητα της συζήτησης αυτής σε διάφορα κράτη-μέλη μας δείχνει ότι έχουν αλλάξει οι όροι θα πρέπει να προσέξουμε ότι μια νέα αποτυχία δεν θα ήταν ε, αποδεκτή. Το τελευταίο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλήλως όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ένωση και την Μεγάλη Βρετανία. Η κυρία Μπερές θέλει να χαιρετήσει και πάλι την εργασία των δύο εισηγητών και τους εύχεται να καταφέρουν να φτάσουν σε μια φιλόδοξη πρόταση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να οθεθεί και το Συμβούλιο σε μια συμφωνία σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σάντερ Ζάντερ Λούμς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι από μια εξαγωγική περιοχή, μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική περιοχή της χώρας μου. Τα θέματα λοιπόν της ε, φορολογικής βάσης και της φορολογίας με ενδιαφέρουν. Και όπως ξέρετε ο διάβολος πολλές φορές είναι στις λεπτομέρειες αυτά τα θέματα. Διότι η κατάσταση και η φορολογική αντιμετώπιση της κάθε επιχείρησης και της κάθε χώρας μπορούν να διαφέρουν. Γι' αυτό θέλει η Κομισιόν να εναρμονίσει από την πίσω πόρτα τη φορολογική βάση. Ξέρουμε τι συνέβη την τελευταία φορά με αυτή την πρόταση. Πήγε στο καλάθι. Είπατε κύριε Τάν ότι η εναρμονισμένη βάση θα φέρει πλέον εκτήματα και απλούστευση. Απλούστευση στα λογιστικά των επιχειρήσεων. Αλλά τι θα γίνει με αυτούς τους φόρους. Όπως ξέρετε, το θέμα είναι πώς δαπανώνται οι φόροι αυτοί από τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, τα έσοδα των επιχειρήσεων που έχουν ε, πολλές έδρες για παράδειγμα, πώς κατανέμονται τα φορολογικά τους έσοδα στα διάφορα κράτη-μέλη όπου δραστηριοποιούνται. Γιατί ξέρετε, το θέμα είναι για το ψητό. Οι χώρες που είναι ανταγωνιστικές ε, και οι οποίες έχουν ε, καταφέρει να είναι ανταγωνιστικές λόγω των μεταρρυθμίσεων που έχουν κάνει, δεν πρέπει να τιμωρηθούν γι' αυτό. Αλλά εδώ προτείνεται ακριβώ μια μεταβίβαση φορολογικών σώδων από τι καλύτερες χώρες στι χειρότερες. Αυτό λοιπόν προτείνεται. Αυτό προσπαθεί η Κομισιόν. Θέλουν βεβαίως αυτή η εναρμόνιση να γίνει σταδιακά. Στην αρχή θα είναι θελοντική υποτίθεται, αλλά τελικά θα γίνει υποχρεωτικό το σύστημα, με βάση καθορισμένα κατόφλια. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί υπέρ αυτού του συστήματος στο Κοινοβούλιο, αλλά θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι είναι προβληματικές αυτές οι προτάσεις. Ένα θέμα που δεν είναι καινούριο. Είναι η μελέτη αντικτύπου. Ο κύριο Λαμασούρη είπε, κανείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει, ούτε καν η Επιτροπή. Κανείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τη πρόταση αυτής να μας δώσει νούμερα για το τι θα συμβεί. Όμως, χρειαζόμαστε μία ανάλυση. Και ε, αυτή η ανάλυση υπάρχει τελικά, διότι η Κομισιόν λέει ότι θα έχει θετικέ επιπτώσει για την οικονομία τη Ένωση η εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Μα τι πάνε Ε, ορισμένοι λένε ότι θα έχει ουσιώδει επιπτώσει. Το είπε και ο κύριο Φέρμπερ. Οι επιπτώσει θα είναι ουσιώδει. Έτσι είπε. Μα είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Είναι δυνατόν ε, να περιγράφουμε τις επιπτώσεις τόσο γενικόλογα χωρίς καθόλου νούμερα. Πώ ακριβώς θα είναι, ούτε καν την περιγράφουμε την κατάσταση που θα προκύψει. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι και όχι τόσο ασαφεί. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση της κατάστασης. Και έχουμε δει μελέτες από τις ε, μεγάλες εταιρείες ε, συμβούλων οι οποίοι έχουν ε, αποτιμήσει τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα κράτη. Και για τα μικρότερα κράτη-μέλη οι προβλέψεις που κάνουν είναι αρνητικές. Ε, λέμε ότι θέλουμε να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις. Συμφωνώ κύριε Τόγκ, αλλά να προσελκύσουμε με φορολογικά κίνητρα τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξέρω αν είναι πάντα η σωστή μέθοδος διότι ακριβώς θα πληρώσουν ε, το κόστος κατόπιν οι χώρες οι οποίες θα έχουν προσελκύσει τις επιχειρήσεις που θα έχουν τα κέρδη. Και δεν τους παραμένει καμία δυνατότητα να συνεχίσουν ε, να ασκούν μία πολιτική φορολογική. Η Μάλτα, για παράδειγμα, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα. 5% για όλους. Γιατί βέβαια το θέμα είναι ποιος θέλει να πάει σε τόσο απομακρυσμένο σημείο της Ένωσης. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι δυνατόν να δώσει κάποια κίνητρα μια χώρα για να προσελκύσει ε, επιχειρήσεις. Όπως και η Ιρλανδία βεβαίως. Αλλά το ερώτημα που τίθεται αν είναι σωστή η πολιτική που ασκεί η Ιρλανδία όταν προσελκύει μόνο με τέτοιου τύπου κίνητρα επιχειρήσεις. και όπως ξέρετε ήδη το 2011 η κλίδα κατανομής των φορολογικών εσόδων ήταν ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Διότι σημαίνει ότι τα μικρότερα κράτη-μέλη δεν θα ωφεληθούν τελικά από μια τέτοια κλίδα κατανομής. Άρα θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι συνάδελφοι από τα μικρότερα κράτη-μέλη. Αυτή η υποτιθέμενη πανάκια νομίζω ότι στην ουσία θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Συζητήσαμε για τη φορολογική βάση, αλλά εδώ ε, τίθεται και το θέμα των συντελεστών. Για τους ίδιους πόρους, όλα όσα δεν έχουν συζητηθεί ακόμη, παρουσιάζουν ακόμη περισσότερες παγίδες. Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί πολύ περισσότερο σε βάθος τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμόνισης, αλλά εναρμόνισης προς όφελος πιανού. Θα αποφεληθούν μόνο τα μεγάλα κράτη-μέλη, όχι όλα τα κράτη-μέλη. Ενώ αντίθετα, ε, εμείς πάντα πιστεύαμε ότι θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να ωφελεί όλους. Άρα στόχος μας πρέπει να είναι βεβαίως τα μικρότερα κράτη-μέλη να έχουν με σωστό τρόπο τη δυνατότητα να παραμείνουν ανταγωνιστικά, να είναι ελκυστικά για τις επιχειρήσεις μέσω της ε, φορολογικής τους πολιτικής. Αυτό που θέλουμε όμως βεβαίως είναι θεμητός, δίκαιος ανταγωνισμός. Αυτή είναι η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ιδιαίτερα λάθος που αυτή η τόσο θεμελιώδη συζήτηση δεν γίνεται όταν συζητάμε ένα, ένα τόσο σημαντικό θέμα. Τώρα πρέπει να πάω ψηφίσω την ίντα, αλλά θα επανέλθω και θα παρακολουθήσω τη συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Well... Ευχαριστώ. Για το CCTV. θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πολ Τάνκ ε, για την εργασία του επί αυτού του θέματος. Ε, σωστά ανέφερε στην έκθεσή του ότι αυτό το ζήτημα είναι ε, ένα από τα λιθαράκια που λείπουν από το νομικό μας οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή. Είναι πολύ σημαντικό η ενοποίηση της φορολογίας να παραμείνει ως βασικό στοιχείο ε, αυτής της πρωτοβουλίας ε, ε, με την ενοποίηση, την τρύπα του transfer pricing και γενικά με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, γι' αυτό και οι δύο εισηγητέ έχουν συνδέσει αυτές τις δύο πρωτοβουλίες και εκθέσεις που αφορούν δύο διαφορετικές οδηγίες. Ένα άλλο θέμα είναι η φορολόγηση του ψηφιακού τομέα. Η ψηφιακή διάσταση θα πρέπει να υπάρχει και στον ορισμό της μόνιμης έδρας. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει γιατί ε, θα πρέπει να ενσωματώσουμε και το ζήτημα της φυσικής παρουσίας ε, μιας εταιρείας που δεν είναι απαραίτητη όταν έχουμε ψηφιακή ε, υπηρεσία. Επίσης, η ιδέα των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών επί της ουσίας και δεδομένης και της αντίστασης διαφόρων κρατών μελών σε όλη αυτή την πρωτοβουλία ε, θεωρώ ότι αποτελεί μια κερκόπορτα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να σκοτώσουμε αυτή την ε, πρωτοβουλία. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να έχουμε ένα όριο, ε, αλλά αναρωτιέμαι πώς αυτό θα λειτουργήσει στην πράξη. Θα, θα έχουν λοιπόν τα κράτη-μέλη ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα άλλο για τις πολυεθνικές. Επίσης η παρακράτηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, αυτό το κόστος, ε, θα πρέπει οι πολυεθνικές να μην χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο μόνο για φορολογικούς λόγους, ε, ο εισηγητής άλλαξε το νούμερο εδώ και αναρωτιέμαι γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο νούμερο. Επίσης, ε, εφόσον ο όλα άλλαξε αυτά τα νούμερα, μπορεί να μας εξηγήσει το σκεπτικό του. Ευχαριστώ πολύ και αντιμονώ για μια περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος. Ευχαριστούμε. Ματ Κάρθη. Υπάρχει και η κυρία Βίρινγκ που θέλει το λόγο πρώτη. Ε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, την, ε, το σχέδιο πρόταση του κυρίου Λαμασούρ που είναι ισορροπημένο και αποτελεί μια καλή βάση συνεργασίας. Να επικεντρωθώ στο γεγονό ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτές τελικά θα υποφεληθούν περισσότερο από το νέο σύστημα. Δεν έχουν την πολυτέλεια να αντιμετωπίσουν 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα πόσο μάλλον τους για να χρησιμοποιήσουν την πιο κερδοφόρα φορολογική πολιτική. Γι' αυτό πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν ίσοι όροι και ίσες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Ο ΚΕΦΕ είναι λοιπόν μια νέα ευκαιρία να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το σύστημα ανταγωνισμού. Επίσης, χαιρετίζω το γεγονός ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το νέο σύστημα εθελοντικά και τους, ε, τις προσκαλώ να το κάνουν. Επίσης, ε, η ΚΕΦΕ θα έχει πολλές, ε, πολλά πλεονεκτήματα παρόλο που θα υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής που είναι απαραίτητη όταν περάσει αυτή η περίοδος θα υπάρχουν σημαντικές εξοικονομήσεις σε διοικητικό κόστος. Πρόκειται λοιπόν ε, τέλος για μια πρόταση η οποία στην ουσία ε, ωφελεί τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Και γι' αυτό είμαι υπέρ και των δύο παρακρατήσεων. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε επίπτωση, καταστροφική επίπτωση στα αφορολογικά έσοδα των ε, κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω λίγο περισσότερα για την πρακτική εφαρμογή. Επίσης, αδειμονώ για άλλες ιδέες και προτάσεις στο ίδιο πλαίσιο. Επιπλέον, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα ε, αν θέλουμε να αλλάξουμε τον προτινόμενο τύπο, την προτινόμενη φόρμουλα. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νέες βιομηχανίες, όμως οι αλλαγές μας θα πρέπει να βασίζονται σε τεκμήρια, συγκεκριμένα αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Η αλλαγή θα πρέπει να λύνει προβλήματα και όχι να δημιουργεί νέα παραθυράκια και κενά. Είναι λοιπόν σημαντικό τα δύο συστήματα, πέραν όλων των άλλων, να τεθούν σε εφαρμογή ταυτόχρονα για να λειτουργήσουν σωστά και να επιτύχουν τους στόχους τους. Για να καταλήξω, και είναι θέμα αντιγωνιστικότητας και ανταγωνισμού. Πρέπει να διατηρήσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών, αλλά ε, αν ε, ασχοληθούμε ε, μόνο με, την, ε, με αυτό δεν θα ασχοληθούμε με την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλήκα. Ευχαριστώ. Και τώρα Μακάρθη. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την εργασία τους επί του σχεδίου έκθεσης. Θα μιλήσω και για τις δύο εκθέσεις, θα δώσω τις απόψεις μας και θα σας πω κάποια από τα ζητήματα που, με που απασχολούν και τους άλλους συναδέλφους από την ΚΟΕ, όπως ε, ο μαθηματικός τύπος. Όσοι είναι υπέρ της φορολογικής επικράτειας και εθνικής κυριαρχίας ε, και της διαφάνειας είμαι κατά οποιασδήποτε τέτοια απόφαση ε, που λαμβάνονται από δημοκρατικά εκλεγμένες ε, που δεν λαμβάνονται από δημοκρατικά εκλεγμένες ε, κυβερνήσεις αλλά από την Κομισιόν. Καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή και αποφυγή από τις πολυεθνικές. και οι τροπολογίες που δίνουν την εξουσία στην Κομισιόν να θεσπίζει φορολογικούς συντελεστές είναι κάποιες που δεν θα υποστηρίξουμε. Ε, φαίνεται ότι ε, τόσο αντάλλαγμα ε, για την εισαγωγή αυτού του συστήματος ε, θα μας δίνεται η δυνατότητα οι πολυεθνικές να μην χρησιμοποιούν τα ευνοϊκά συστήματα. Η ΚΕΒΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μας ε, θέτει ενώπιον του κινδύνου να περιχαρακωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να απομονωθεί από τις άλλες χώρες και να υπάρχει μια επιδείνωση ε, τις τάσεις ε, να πηγαίνουν ε, τα κέρδη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολύ ελάχιστα μέτρα που προτείνονται για να αποφευχθεί αυτό μέσα από τις προτάσεις για τον έλεγχο των ξένων εταιριών και οποιαδήποτε πρόταση για το υφερολογία ξένου εισοδήματος. Ε, η πρόταση της Κομισιόν αναφέρει ότι πρέπει κανείς να είναι φορολογούμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής εν μέρη έχει αναφέρει αυτό το θέμα στην έκθεση του για το CCTB. Ε, όμως, ε, τι γίνεται με την κοινή ιδιοκτησία και έλεγχο των εταιριών. Επίσης, ενοποιημένοι λογαριασμοί των εταιριών είναι ένα θέμα που θέτει διάφορα ζητήματα. Ε, δεν υπάρχει κάποια συνέπεια στον τρόπο που υπολογίζονται οι φόροι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και καλό θα ήταν η έκθεση να κάνει κάτι γι' αυτό. Την επόμενη εβδομάδα η ομάδα μας ε, θα δημοσιεύσει μία μελέτη για τις επιπτώσεις του CCTB στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών. Ακόμα είναι υπό προετοιμασία και δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει, όμως ε, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση των φορολογικών εσόδων από αυτή την ενοποίηση και όχι ε, αυτή η εξοικονόμηση που θέλουμε. Ε, μέσω της ενοποίησης, ε, αν η ενοποίηση γίνει από μόνη της και δεν υπάρχει σωστή κατανομή και ένα σύστημα ενιαίο, ε, δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το καναδικό σύστημα, για παράδειγμα, για την κατανομή των πολίσεων των εργοδοτών είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί αξιολογεί την αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία του ενεργητικού με σωστό τρόπο. Η CCTV, λοιπόν, ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ε, για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να έχουν τα μέγιστα αποτελέσματα από τα ε, συστήματα φοροδιαφυγής. Υπάρχουν επίσης αμερικανικές ε, πολυεθνικές ε, που δρούν σε αυτή την κατεύθυνση και, καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι πόροι που μας δίνονται για να έχουμε πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα ώστε να κάνουμε μία ανάλυση. Ιδάλλως θα είναι ανεύθυνο οποιοδήποτε βήμα ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Sent the written intervention of for the record. Ε, έχουμε και την παρέμβαση της Eva για τα πρακτικά. Μπορώ να σας διαβάσω αν το επιθυμείτε. If green, uh, um, okay, so. Α, θέλετε, όχι. Ο Μάρκο Βάλλη τότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία των δύο εισηγητών, γιατί είναι στην ίδια γραμμή με τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή Τάξε και Panama Papers. Μετά από τα, βέβαια τα στοιχεία θα δείξουν όταν θα ψηφιστούν οι νομοθετικές διατάξεις, θα δούμε αν ε, τελικά θα τεθούν σε εφαρμογή. Σε αυτό το είδος προτάσεις συχνά βρίσκουμε συνένεση και μετά συμβαίνει κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να εξηγήσουμε στο κοινό όπως έγινε με το country by country reporting ε, πριν το καλοκαίρι, όπου η πρόταση του Κοινοβουλίου βούλιαξε. Όσον αφορά το κείμενο λοιπόν, με βρίσκει σύμφωνο αν και εμείς σε σχέση με το κείμενο της Κομισιόν, όπως και οι συγητές, δεν στηρίζουμε την ε, προσέγγιση σε δύο φάσεις, γιατί πιστεύουμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή φορολογική βάση που θα είναι ενοποιημένη ταυτόχρονα. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια ολοκληρωμένη πρόταση γρήγορα και να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε όσο γίνεται περισσότερη πίεση στο Συμβούλιο, ώστε ακριβώς τα κράτη να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις τους. Όσον αφορά την έκθεση του Πολ, πιστεύω ότι η μείωση του κατοφλίου είναι κάτι το δίκαιο και τα 750 εκατομμύρια είναι υπερβολικά. Η πρότασή σας μας βρίσκει σύμφωνος. Και θα μπορούσαμε ίσως κάπως να συζητήσουμε για το νούμερο, αλλά ε, είναι λογικό το να μειώσουμε αυτό το κατόφλι και συμφωνούμε και για την φορολόγηση ενός ελάχιστου ε, ποσοστού, ε, ώστε να μην υπάρξει ανταγωνισμός προς τα κάτω. πρέπει να δούμε ποιο είναι το σωστό ποσοστό θα πρέπει από τεχνικής άποψης να το διευκρινίσουμε. Τώρα, η σούπερ μείωση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι ένα νέο σύστημα φορολογικών κινήτρων που ε, αντικαθιστά το patent box και κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλό να μην δημιουργήσουμε ένα άλλο σύστημα κινήτρων που να αντικαθιστά το patent box και για την πρόταση των δύο για τμήμα της φορολογικής βάσης που θα εντάσσεται στον κοινοτικό προπολογισμό θα πρέπει αυτό να αφαιρεθεί από τις εθνικές συμβολές και αυτό θα διευκολύνει και όλα στην αποδοχή από πολλές κατρομελών μιας τέτοιας πρότασης. Αυτές είναι οι βασικές μας παρατηρήσεις, αλλά μπούμε στην ουσία όταν θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Μπάρμπαρα Κάπελα. Α, εσείς θα πάρετε το λόγο. Ναι, η κυρία Κάπελ απουσιάζει και ζητά συγγνώμη. Μπορώ να πάρω το λόγο στο, στη θέση της, κύριε Πρόεδρε. Oui. Yeah, yeah, of ναι, ναι, βεβαίως. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να συγχαρώ του δύο εισηγητέ ε, για την ποιότητα των εκθέσεών τους ε, και τον κύριο Τάν και τον κύριο Λαμασούρ για αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα όπου τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παιδεύονται εδώ και χρόνια. Το διαπιστώσαμε μετά από το σκάνδαλο το LuxLeaks. Το διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα γιατί πρόκειται για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που χάνουμε ε, και είναι φυσικά παράδεκτο αυτό. Μια παρατήρηση για τον κύριο Λαμασούρ και μια ερώτηση. Ε, πρώτη, νομίζω πως απαντήσατε στις ανησυχίες μας που σχετίζονται με το γαλλικό ε, σύνταγμα της ισότητας απέναντι στους φόρους. Εάν καταργηθεί το κατόφλι, νομίζω πως θα απαντήσουμε σε αυτό το θέμα των δύο φορολογικών καθεστώτων στην διαχώρα. Πιστεύω πως είναι κάτι λοιπόν που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα ε, υπάρχει το θέμα γιατί στη Γαλλία έχουμε την φορολογική διάταξη για τις ε, φοροαπαλλαγές όσον αφορά την έρευνα. Αυτό λοιπόν εδώ μήπως αμφισβητήσει την ε, δυνατότητα απαλλαγής, φόρο απαλλαγής μάλλον των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ωραία. Τώρα έχουμε το Catch the Eye. Ο κύριος Χαρέγγιρη του Όντο, πρώτος έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ότι όντως έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και η εργασία των δύο εισηγητών, Τάγκα και Λαμασούρα, είναι εξαιρετικά σημαντική. Θεσπίζονται όμως κάποιες ε, βασικές αντιρρήσεις, ενστάσεις ε, σε αυτή. παραβάσεις που ήταν βασικά κατά. Από τη μια πλευρά έχουμε να κάνουμε τη φορολογική αρμοδιότητα. Ορισμένε περιφέρειες, η κράτη ευρωπαϊκά, χρειάζονται να μπορούν να παίζουν με την φορολογία για να είναι ανταγωνιστικές ή ανταγωνιστικά. Ή μιλάμε για φορολογική κυριαρχία. Εγώ πιστεύω πως οι συνάδελφοι που παρεμβαίνουν υπερασπιζόμενοι την φορολογική κυριαρχία ή την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών ξεχνούν πως είμαστε σε μια νέα αγορά και ότι δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι ε, πληρώνουν ή δεν πληρώνουν οι πολυεθνικές, ε, πληρώνουν σε μια χώρα προς όφελος των άλλων. Για να αποφύγουμε λοιπόν τα rulings, να αποφύγουμε την τεχνητή μεταφορά κερδών, ε, ένα σωρό αδικίες δηλαδή φορολογικές και βλάβες εις βάρος των κρατών πρέπει να δράσουμε. Και γι' αυτό το λόγο το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη γνώμη μου σε αυτήν εδώ την έκθεση θα μπορούσε να δείξει, να, να, μάλλον μόνο να συμβουλέψει γιατί δεν συνομοθετούμε εδώ, όμως πρέπει να δώσουμε τη γνώμη μας και η γνώμη μας πρέπει, θα πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση και να ενίσχυση συγγνώμη, της, της οδηγίας και όχι να αποδυναμωθούν τα μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν στο Συμβούλιο. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει με ομοφωνία και θα ακούσει μόνο τη γνώμη μας. Άρα λοιπόν πιστεύω πως η γνώμη μας θα πρέπει να είναι πολύ σημαντική και πολύ ε, ξεκάθαρη και γι' αυτό θέλω να δείξω την ικανοποίησή μου γιατί πολλές από τις τροπολογίες τόσο του κυρίου Λαμασού όσο και του κυρίου Τάγκ ε, ε, είναι πολύ ειδικά, ειδικές, ας πούμε μείωση κατοφλίου στα 40 εκατομμύρια σε σχέση με την πρόταση επίσης για το φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη συμπερίληψή του. Λοιπόν, εδώ η ιδέα της ε, μετατροπής ενός τμήματος της φορολογικής βάσης σε ίδιο πόρο ε, για τον προπολογισμό της Ένωσης είναι σημαντικές ιδέες. Να τελειώσω με δύο, με μου, ε, δικούς μου προβληματισμούς. Πρώτον, η μείωση της αποζημίωσης που προβλέπεται για την ε, σαπόλης ε, τις ζημιές ε, λόγω της δημιουργίας της φορολογικής βάσης. Ένα δις έχει υπολογίσει η Κομισιόν αυτή την αποζημίωση, γιατί η Κομισιόν υπολογίζοντας όλους αυτούς τους μηχανισμούς μείωσης, έκπτωσης κτλ που ισχύουν σε όλες τις χώρες έχει φτιάξει ένα σύστημα τόσο μεγάλο γενίκευση όπου ο αντίκτυπο θα είναι σημαντικό όσον αφορά αυτή τη μεταρρύθμιση. Γι' αυτό και μου άρεσε αυτή η ιδέα του κυρίου Λαμασούρ να φτιάξουμε ένα προσωρινό ταμείο αποζημίωση για τα κράτη που θα χάσουν από αυτή την υπόθεση. Και για τέλο, ένα δεύτερο προβληματισμό σε σχέση με το σύστημα ενοποίηση. Γιατί ε, ίσως ε, κύριε Λαμασούρ να υποβάλω μια τροπολογία γιατί δεν, νομίζω πως δεν έχετε ε, λάβει επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι οι συγκρούσεις όσον αφορά την καταβολή των φόρων θα επιτρέψει στις, στις εταιρείε να επιτρέψουν τη δικαιοδοσία στην οποία θα υποβάλουν αυτές τις διαφορές και συγκρούσεις. Άρα λοιπόν, επειδή θα υπάρξουν προβλήματα ανάμεσα στα κράτη, θα πρέπει να ορίσουμε μια πιο αντικειμενική βάση καταχώρησης της δικαιοδοσίας προς το αρμόδιο κάθε φορά κράτος, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κράτος και την, την ενοποιημένη φορολογική βάση. Να δείξουμε δηλαδή ε, και να επαναλάβω άλλη μια φορά πως το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει μια γνωμοδότηση κοινή και ισχυρή σε μια συζήτηση που όχι μόνο είναι επίγουσα, αλλά είναι και απαραίτητη ώστε να επικρατήσει φορολογική δικαιοσύνη. Ο Μπέρντ Ευχαριστώ, μια τόσο θεμελιώδης μεταρρύθμιση όπως αυτή που προτείνουν οι δύο εκθέσεις έχει πολλά υπέρ και κατά. Ορισμένα ήδη προαναφέρθηκαν. Και στην ομάδα μας υπάρχουν ε, διχογνωμίες. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση θετικά, ίσως πιο θετικά από ό,τι φάνηκε από αυτά που είπε ο συνάδελφος Ζάντερ αν και μπορώ να υποστηρίξω πολλά από τα επιχειρηματά του. Να τονίσω. Οι δύο προσπάθειες αυτές βεβαίως ε, συνδυάζονται, αλλά ίσως καλύτερα να εφαρμοστούν ε, η μία ε, μετά την άλλη. Θα μας επιτρέψουν να λύσουμε πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουμε στην Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι η φορολογική βάση πολλές φορές δεν είναι εκεί που λαμβάνει η χώρα η οικονομική δραστηριότητα και συνειδητά κάποια κράτη-μέλη με, χαμηλότερους, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές προσπαθούν να προσελκύσουν ε, φορολογική βάση που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε άλλη χώρα. Επίσης υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν διαμεθοριακά και έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις διαφορές μεταξύ φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών με τρόπο που δεν είναι λογικός. Ένα άλλο πρόβλημα που θα λύσουμε είναι ότι θα έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα τα οποία θα μπορούσαμε τουλάχιστον εν μέρη να δαπανίσουμε, ούτω ώστε τα μικρότερα κράτη-μέλη που μπορεί να θυγούν από αυτή την αλλαγή τη φορολογική βάση να αντισταθμίσουν αυτέ τι απώλειε. Όμω, εφόσον θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή και θεωρούμε ότι είναι άδικη η φορολογική η κατανομή της φορολογικής βάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να την ε, δεχτούμε. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτή την προσπάθεια προσέλκυσης με τεχνητό τρόπο φορολογικής βάσης. Έτσι θα λύσουμε πολλά συστημικά προβλήματα. Αλλά αν η πρόταση αυτή συνδυαστεί με θέματα που είναι άσχετα, για παράδειγμα ελάχιστος φορολογικός συντελεστής, τότε για μένα και πολλούς άλλους στο, ECR θα ε, παραβιαστεί μια κόκκινη γραμμή κάτι που θα σήμαινε ότι θα είμαστε κατά γιατί ο ελάχιστος φορολογικός δελεστής δεν έχει κανένα ρόλο σε μια τέτοια πρόταση. Εάν η φορολογική βάση καθοριστεί έτσι στα πλαίσια του CCTB, ούτως ώστε η οικονομική δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα στην σωστή δικαιοδοσία, δεν υπάρχει πια καμία αιτιολόγηση να πούμε εμείς ε, με τι συντελεστέ θα φορολογήσει ε, την οικονομική αυτή δραστηριότητα. Αυτό είναι η δική του πλέον φορολογική βάση. Δεν είναι ξένη φορολογική βάση την οποία έχει προσελκύσει με τεχνάσματα. Για μένα λοιπόν θα ήταν απαράδεκτη ε, μια προσπάθεια επιβολής ελάχιστου φορολογικού συντελεστή. Επίσης η πρόταση ότι το CCTV, CCCTV, ο εταιρικός φόρος, πρέπει να αξιοποιηθεί για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα της Ένωσης. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αν θέλουμε να υπάρξει μια επιτυχής πρόταση μεταρρύθμισης της φορολογικής βάσης, δεν πρέπει να το συνδυάσουμε με άλλα περιεχόμενα. Δεν πρέπει με, από το παράθυρο να βάλουμε άλλα θέματα στην εξέταση του θέματος αυτού γιατί θα μειώσουν την αποτελεσματικότητά του. Αυτές λοιπόν είναι δύο κόκκινες γραμμές που για μένα μπορούν να αποτελέσουν λόγο να καταψηφίσουν το CCCTB. Κατά τη γνώμη μου, όπως είπα προηγουμένως, και όπως έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν καλύτερα να διαχωρίσουμε τις ε, δύο αυτές προτάσεις. Η ενιαία βάση να είναι η πρώτη πρόταση και η ενοποιημένη ενιαία βάση να έρθει αργότερα. Γιατί μόνο και μόνο ο ορισμός του τι σημαίνει κέρδος θα μας επιτρέψει να κάνουμε μετά την μελέτη των επιπτώσεων που ανέφεραν ορισμένοι. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε τι οικονομικές και φορολογικές επιπτώσεις έχει το θέμα αυτό. Εάν καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό του τι σημαίνει φορολόγηση κέρδος, τότε θα έχουμε ήδη μια βάση. Εάν επιδιώξουμε περισσότερα, τότε θα αυξηθούν και οι αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις που θα υπάρξουν αν επιχειρήσουμε να τις περάσουμε για το δύο μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Σβέν, θα μας παρουσιάσετε την πρόταση της ε, ομάδας σας. Παρακαλώ. Ναι, πήγε ταχύτερα από ό,τι περίμενα συζήτηση. Η Εύα Ζολή ήταν η δεν μπορεί να παρευρεθεί. Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο που μου έδωσε. Γενικά χαιρετίζουμε τη νέα όθηση που δόθηκε για τις δύο αυτές προτάσεις. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε το ότι η Κομισιόν παρουσιάζει την ενοποιημένη βάση μαζί με την κοινή βάση, την ενιαία βάση. Χαιρετίζουμε τις προτάσεις Ταν και Λαμασούρ, ιδιαίτερα τη σαφή πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν παράλληλα τις δύο προτάσεις, ταυτόχρονα. Οι τροπολογίες είναι πολύ θετικές, γιατί δεν ήταν σαφές ε, στην πρόταση της Επιτροπής εάν και κατά πόσο τα δύο θέματα αυτά θα συζητηθούν σε δύο διαφορετικές φάσεις ή ταυτόχρονα. Καλωσορίζουμε επίσης το ότι οι εισηγητές διατηρούν τη βασική αρχή της πρότασης της Κομισιόν. Δηλαδή ότι το νέο σύστημα αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τις μεγαλύτερες εταιρείε. Κάτι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη προτείνει από το 2012. Πρέπει οι μεγάλες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν δεσμευτικά με το σύστημα αυτό. Διότι αν γινόταν με θελούσιο τρόπο θα είχαμε 29 τρόπους φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αντί να αντικαταστήσουμε τα 28 συστήματα με ένα κοινό σύστημα. Σημειώνουμε ότι τα σχέδια εκθέσεων είναι ακόμη πιο φιλόδοξα. Θέλουν αυτό το νέο σύστημα να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις. Προσβλέπουμε στη συζήτηση των υπέρ και κατά της πρότασης αυτής. Στηρίζουμε τις απόψεις των εισηγητών ότι ένα τμήμα των φορολογικών εσόδων από την κοινή ενιαία βάση θα πρέπει να είναι ίδιος πόρος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Σύμφωνα με τις προτάσεις ε, του, της ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους, αλλά αυτή η πρόταση πρέπει να είναι πιο αναλυτική ο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στου ε, ενωσιακού ίδιου πόρου πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Ω πράσινοι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα εναρμονισμένο και δεσμευτικό ορισμός της μόνιμη εγκατάσταση. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τι προτάσει των συγητών για έναν ακριβή και δεσμευτικό ορισμό των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρεί μια πολυεθνική για να αποδείξει ότι βασίζεται στην αλφα χώρα και θα έπρεπε να ισχύουν τα κριτήρια αυτά και για τη μη ηλική ψηφιακή δραστηριότητα. Ένα τέτοιο δεσμευτικό ορισμό θα απέφυγε καταστάσει όπω αυτέ που είδαμε πρόσφατα στη Γαλλία, όπου ένα δικαστήριο αποφάσισε ότι η εταιρεία Google δεν είχε μόνιμη εγκατάσταση στη Γαλλία, άρα δεν έπρεπε να φορολογηθεί στη Γαλλία. Συμφωνούμε να αρχίσουν να ισχύουν αυτές τις προτάσεις το 2020. Τώρα, σχόλια για την έκθεση ΤΑΝ. Καλωσορίζουμε την εναρμονισμένη, τον εναρμονισμένο ορισμό της ε, μυστικότητας και της ε, ε, ενωσιακής δικαιοδοσίας πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω τα κριτήρια στο σημείο 21. Η διατύπωση όμως δεν πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες που ακόμη δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για φορολογικά θέματα. Ως πράσινοι πιστεύουμε επιπλέον ότι το CCCTB θα έπρεπε να εισαχθεί παράλληλα με τον ελάχιστο εταιρικό συντελεστή φορολόγηση. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τι προτάσεις του συγητή. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μέχρι την 1η Πρώτου 19 νομοθετικές προτάσεις για έναν ελάχιστο αποτελεσματικό ε, εταιρικό φόρο 18% συντελεστή δηλαδή. Ο συντελεστής αυτός βέβαια θα πρέπει να συζητηθεί. Αλλά είναι σωστή γενικά η πρόταση. Η εισαγωγή μιας κοινή εταιρική φορολογικής βάσης είναι μόνο το πρώτο βήμα για να αντιμετωπιστεί η φόρο αποφυγή και ε, το φορολογικό dumping. Πρέπει αυτή η βάση να συνδυαστεί λοιπόν με έναν ελάχιστο εταιρικό συντελεστή για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός ε, συντελεστών. Για την έκθεση Λαμασούρο, ο εισηγητής ζητάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια αποτίμηση της πρότασής CTB κάθε χρόνο. Συμφωνούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρω για την εφαρμογή και λειτουργία αυτού του νέου συστήματο, γιατί δεν θα έπρεπε να αναλάβει η Επιτροπή αυτή την αποτίμηση και να την ε, ε, αποστέλει πλήρως στους ε, βουλευτές. Έχουμε αμφιβολίες για το προσωρινό Ταμείο Αποζημίωσης για να αντισταθμιστούν, αντισταθμιστούν οι ζημίες. Από την εισαγωγή του νέου συστήματος καταλαβαίνουμε ότι θα διευκόλυνε την εισαγωγή του και θα έπιθε κάποιους απρόθυμους. Θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου δεν είναι η καλύτερη λύση. Και η κατάργησή του ε, αργότερα δεν θα είναι εύκολη. Τέλος, σημειώνουμε ότι αν δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση, οι εισηγητές προτείνουν να εγκριθεί μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να περάσει από το Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μας υπάρχει και άλλη λύση. Προτείνουμε η Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση που να βασίζεται στο άρθρο 116 της συνθήκης, δηλαδή την αντιμετώπιση της τρέβλωσης του δανεισμού στην ε, ενιαία αγορά, κάτι που θα επέτρεπε να εγκριθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία και όχι ομοφωνία. Αυτό θα μας ε, βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ότι ορισμένοι αποφεύγουν την πρόταση αυτή για, να μην, για, για λόγους, δηλαδή για να έχουν κέρδος. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, κύριος Αρτοβαχίλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, χαιρετίζουμε τις ε, θετικές παρατηρήσεις και τα σχόλια που εξέφρασαν οι εισηγητές, οι σκιώδες εισηγητές και οι διάφοροι ομιλητές. Φαίνεται ότι γενικά υπάρχει υποστήριξη εκτεταμένη παρόλο που υπάρχουν παρατηρήσεις για συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν διάφορα σημεία που θα ήθελα να θέσω. Η ψηφιοποίηση καταρχάς της οικονομίας και τα ζητήματα που αφορούν στον τρόπο φορολόγησης αυτών των υπηρεσιών και πώς καταβάλλεται αυτός ο φόρος. Αυτά είναι ζητήματα που οπωσδήποτε γερονται μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό χαιρετίζουμε στις 15 Σεπτεμβρίου τη συζήτηση που θα γίνει με πρωτοβουλία της Εστονικής Προεδρίας στο Ταλίν. Γιατί χρειάζεται μια ενδελεχής ανάλυση του, των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτόν το τομέα και του τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να βελτιώσουμε την πρόταση για την κοινή βάση και την βάση για την ΚΕΠΦΕ Όμως, αυτό που πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει είναι να εργαστούμε ώστε να υπάρχει μια συντονισμένη προσέγγιση και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την πλευρά των τρίτων χωρών οι, οποίοι θα, οι οποίες θα έρθουν στο τραπέζι για να συζητήσουν το πώς θα βελτιώσουμε την φορολόγηση χωρίς να υπάρχει πρόθεση τιμωρίας ή διπλή φορολόγηση ή υψηλότερη φορολόγηση των ευρωπαϊκών εταιριών και των εταιριών που δρούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια βέβαια ανησυχούν ιδιαίτερα για θέματα επικουρικότητας αναφέρθηκε το θέμα της εθνικής ε, κυριαρχίας ε, και είναι δύσκολο κανείς εύκολα να αποδεκτεί κάτι που παραβιάζει τις ε, αρμοδιότητες και εξουσίες του παρόλο που ενδεχομένως τελικά να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Το κατόπιλο που προτείνει η Κομισιόν είναι 750 εκατομμύρια όμως ξεκάθαρα φαίνεται πως ε, το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους συζητητές και τους άλλους ενδιαφερόμενους αλλά φυσικά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν λόγο για το κατά πόσο θέλουν να προχωρήσουν, πόσο μακριά θέλουν να πάνε. Για την έλλειψη δεδομένων και το πώς αναλύεται ναι. όπως αναλύονται τα, φορολογικά, τα έσοδα στον προϋπολογισμό, τα δημοσιονομικά έσοδα. Ε, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου από την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας. Παρακαλώ, σύντομα αλλά το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι η κυρία Κονέτσνο από την Ταξούντ. Να διευκρινίσω ένα θέμα που έχει συζητηθεί. Μαζί με την πρόταση, η Κομισιόν έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων και θα δημοσιεύσει με ανοιχτό και διαφανή τρόπο όλα τα δεδομένα που προέρχονται από το modeling και όλες τις άλλες μελέτες που έχει διεξαγάγει. Φυσικά το impact assessment είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις και φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, δηλαδή έσοδα, ανάπτυξη. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε επίπεδο κρατών μελών ως προς τη χρήση μοντέλων και την ανάλυση των επιπτώσεων, ε, καλό θα είναι, αν θέλουν τα κρατη να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς. Ευχαριστώ. Να πάμε πίσω στους εισηγητές. Ο καθένας από δύο λεπτά. Αλλά αλλάζουμε και τη σειρά. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεισέφεραν στη συζήτηση και τους σκιώδες και τους υπόλοιπους. Φυσικά υπάρχουν διαφορές ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες, καμιά φορά οι διαφορές είναι μεγάλες, όμως γενικά φαίνεται ότι όλοι εκτός από τον Μπέρντ Λούκε που έχει διαφορετική προσέγγιση, ε, όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι πρέπει να είναι οι δύο προτάσεις συνδεδεμένες. Ο κύριος Λούκε ε, ε, και άλλοι είπαν ότι καλό είναι να αδράξουμε την ευκαιρία για να φορολογήσουμε την ψηφιακή οικονομία. Επίσης, η φόρμουλα που προτείνεται για να ληφθεί υπόψη η ψηφιακή δραστηριότητα στην ενοποίηση είναι κάτι που υπάρχει ήδη σε κάποια κράτη-μέλη. Επιμένω στο γεγονό ότι παρά τους φόβους που έχουν εκφραστεί δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος λόγος. Το σύστημα που προτείνουμε να θεωρείται ότι ε, έχει προνομιακή μεταχείριση για κάποιες χώρες σε σχέση με άλλες. Η κυρία Ζολή είναι λίγο εχθρική, όμως όλοι οι υπόλοιποι είναι υπέρ αυτού στα μέτρα που προτάθηκε και μακροπρόθεσμα, από τη δική μου άποψη, ε, θα υπάρχουν και πολιτικές διαφωνίες γι' αυτό, οι μικρές χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την φορολογία των κερδών για να προσελκύσουν οικονομική δραστηριότητα θα μπορούν να το κάνουν με τους συντελεστές. Επειδή είναι μικρές, ε, θέλουν με τους συντελεστές να προσελκύσουν φόρους που δεν ανταποκρίνονται ε, στην οικονομική δραστηριότητα που υπάρχει σε αυτές. Με το LuxLeaks αυτά αποκαλύφθηκαν και θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος. Πρέπει επίσης να πω ότι όλοι συμφωνούν πως πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να προσέξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα και μόνο σύστημα για όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με μια διαδικασία σταδιακή, σαν αυτή που είπε ο Μάρκους ε, Φέρμπερ, ένα phasing in. Αυτό θα το δούμε. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα ήταν αυτή που είχε να κάνει με το θέμα της δικαιοδοσίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν 27 διαφορετικές ερμηνείες της νομοθεσίας από τα διάφορα εθνικά δικαστήρια. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία ερμηνεία για να μην φτάνουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τέλος. για το ιδιαίτερα γαλλικό σύστημα για το φόρο της έρευνας ε, να πω ότι και στην ίδια την Κομισιόν αυτό το ε, ανάφερε και η Επιτροπή της Γαλλικής Γερουσίας, το ε, γαλλικό σύστημα δεν έχει να κάνει με τη φορολογική ε, βάση, αλλά με την κάλυψη της φορολογίας που δεν είναι στα ίδια πλαίσια και είναι λογικό κάποιες χώρες με τις επιστροφές να στρεβλώνουν το πνεύμα της οδηγίας. Ε, αυτό βέβαια, εάν το γαλλικό σύστημα δηλαδή ε, φανεί ότι είναι το καλύτερο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να πατάξουμε τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ο Πολ Πάνκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ επικοδομητική η συζήτηση σήμερα. Υπάρχουν ε, δυνατότητα να σχηματίσουμε μια σταθερή και ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μέσα από τις συζητήσεις και από τα θέματα που ε, ε, ε γύρατε όλοι οι συνάδελφοι. Πρώτον, οι φοροαπαλλαγές για έρευνα και ανάπτυξη είναι αυτό κομμάτι της σύγχρονης οικονομίας όπου βλέπουμε ίση μεταχείριση των ε, χρεών και του, των ε, περιουσιακών ε, στοιχείων. Πρέπει αυτό να δούμε, πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά όλα αυτά τα, όλα, όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να είμαστε ρεαλιστές και μια γενική φύσης παρατηρήση. Αν θέλουμε αυτή η θέση να ε, ληφθεί υπόψη θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και όσον αφορά τα, ε, τα φορολογικά έσοδα, κάθε χώρα φοβάται μήπως μειωθούν τα φορολογικά έσοδα. Αυτό είναι απίθανο, αλλά είναι ένα δεχόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί είναι σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε την μετάβαση. Η Κομισιόν υποβάλλει μια πρόταση για μετάβαση από τα 2C στα 3C. Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εφόσον πρόκειται για μεγάλη μεταρρύθμιση, μήπως θα πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή του συστήματος. Κάτι επίσης που ανέφερε ο Μάρκος Φέρμπερ, η δική μου άποψη είναι ότι ένα ταμείο αποζημίωσης θα βοηθήσει επίσης αυτή τη μεταβάση, την την μετάβαση μάλλον. Θα είναι πολύ δίκαιο και καλό να βοηθηθεί αυτή η μετάβαση. Ώστε να αντιμετωπιστούν οι μη αναμενόμενες συνέπειες. Ταυτόχρονα πρότεινα εγώ χαμηλότερο καταφύγει γιατί θέλουμε αυτό το σύστημα να ισχύσει όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες αλλά για όλες τις εταιρείες που θα ωφεληθούν από ένα ενιαίο σύστημα. Θέλουμε να εφαρμοστεί λοιπόν σε όλες τις εταιρείες αλλά αυτό παίρνει χρόνο. Γι' αυτό είπαμε να μειωθεί το κατόφλι σε δύο φάσεις. Υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ο Μακάρθι είπε σωστά ότι αν θέλουμε να έχουμε ομοιόμορφη φορολογία θα πρέπει τελικά να καθιερωθεί και παγκοσμίω. Και νομίζω πως η Ευρώπη έχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία να θεσπίσει τα στάνταρ για την ε, φορολογία εταιριών παγκοσμίω. Η Αμερική του Τραμπ προχωρά στην αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό θα έχουμε εμεί τη μοναδική ευκαιρία να θεσπίσουμε προδιαγραφέ για τον εξυγχρονισμό του συστήματο φορολογία εταιριών και την κατάργηση δυνατοτήτων για μετακίνηση κερδών και ε, σχεδιασμό, φορολογικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τη, τι γίνεται στις τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης. Και αυτή η συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να γίνει δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις σχέσεις εκτός Ένωσης αλλά και εντός Ένωσης. Δεν χρειάζεται να έχουμε 27 διαφορετικές ερμηνείες των κρατών μελών, θα πρέπει να έχουμε μια κοινή ερμηνεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και ε, θα περιμένω και τις ε, περαιτέρω συζητήσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Το χρονοδιάγραμμα είναι η κατάθεση τροπολογιών προβλέπεται για τη CCTB στις 25 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα για τη CCCTB 26 Σεπτεμβρίου. Ανταλλαγή απόψεων θα έχουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια στις 10 Οκτωβρίου. Ε, εξέταση των τροπολογιών στις 6 Νοεμβρίου με την ΕΚΟΝ στις 4, 4 Δεκεμβρίου και ε, Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 18, αν είναι δυνατόν. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Ήταν πολύ πλούσια και σημαντική ανταλλαγή απόψεων για ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα για τη φορολογία και για την ε, Ένωση των κεφαλαιοχωρών. Κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών.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 Μία για τις ε, γραμμές, τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να διεξαχθεί οπωσδήποτε τώρα. Για τη δεύτερη ψηφοφορία συνεχίζεται η συζήτηση για μια σειρά θέματα, προφορικές τροπολογίες που μόλις υπευλήθησαν. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, ίσως προτείνει ο εισηγητής να ψηφίσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Αν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Αλλιώς θα ψηφίσουμε και για τις δύο εκθέσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαδικασία του προπολογισμού είναι πάντα λίγο κομική. Πρέπει να υποβάλουμε την πρόταση του σχεδίου έκθεσης τον Ιούλιο γιατί πρέπει να περιμένουμε την πρόταση του Συμβουλίου αλλά πρέπει αμέσως να ψηφίσουμε ε, στην πρώτη συνεδρίαση του Ε, είναι λοιπόν Έγινε λοιπόν εχθές μία συνάντηση των σκιωδών και υπήρξε μια σειρά τροπολογιών συμβιβαστικών ε, για ε, τις φορολογικές βάσεις και ενώ υπήρχε ε, τελικά η συμφωνία ότι θα γίνει η ψηφοφορία. Τώρα έμαθα ότι μια ομάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και δεν έχουν επιληθεί και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Όμως έχουμε τις προθεσμίες και αν δεν το καταφέρουμε να τις στηρίσουμε μέχρι αύριο τουλάχιστον ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και την σωστή διαδικασία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν προτείνω να ε, μην ψηφιστεί τώρα για να ληφθούν τα ανοιχτά ζητήματα. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι τεχνικά ο εισηγητής ζήτησε για αναβολή. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ψηφίσουμε μόνο επί των κονδυλίων του προπολογισμού. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Μήπως να επιχειρήσετε σε κάποιο άλλο μηχάνημα. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία για να ψηφίσουμε και μετά θα συμπολογίσουμε και όσους δεν έχουν μαζί τις κάρτες τους. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας. Και θα προσθέσουμε μία ψήφο ΕΛΚ μόνο, μάλιστα. Εντάξει, η ψήφος ε, των σοσιαλιστών, εντάξει, τώρα καταμετρήθηκε. Ωραία. Τροπολογία οίκων 66-14. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται έκον 6601 και 6625 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται έκον 6612 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έκον 6613 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έκον 6627 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 6617 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 6602 11 και 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Επί της 6606 υπάρχει μια προφορική τροπολογία των πρασίνων να μετακινηθούν 100.000 ευρώ στο αποθεματικό αν εγκριθεί το αρχικό κείμενο πίπτη υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική ορολογία Ωραία, ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66-19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66-15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66-18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66-28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66-05 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 66-05 άρχεται. πέρας εγκρίνεται 66-16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66-08 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, εγκρίνεται συγγνώμη 66 0, 66-07, 66-23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6624 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6604 και 09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6603 και 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6610 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται 42 λοιπόν υπέρ, 7 ε, κατά 5 αποχές εγκρίνεται και συγχαίρουμε τον εισηγητή. Okay, now we move to the next point in the agenda. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημέρης της διάταξης. Πού είναι? το προληπτικό πλαίσιο για την ανεδιάφρωση η δεύτερη ευκαιρία και η διαδικασία για την αφαιρεγγιότητα και την απαλλαγή από τα χρέη. Εισηγητής Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν. Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Πού είναι ο εισηγητής? Θα το βλέπω. Maybe we have been too shocked. Μήπως ε, πήγαμε πολύ γρήγορα την ψηφοφορία και δεν έχει έρθει ακόμη. Ωραία, μια σύντομη διακοπή γιατί έρχεται ο εισηγητής. Okay, short suspension. Λοιπόν, μια σύντομη διακοπή. Uh, λοιπόν, μία που είναι εδώ εισηγητής. Εξάλλου δεν έφταιγε γιατί τελείωσε ταχύτερα η ψηφοφορία. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ήδη παρουσίασα το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν θα, μυρίσω, δεν σφαγιάσω τη γλώσσα του Δάντη, αλλά θα μυρίσω στα ισπανικά και θα σφαγιάσω τη γλώσσα του Θερβάντες. Χαίρομαι που έχω δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας για το πώς να βελτιώσουμε ένα κείμενο που είναι θεμελιώδες κατά τη γνώμη μου για το μέλλον της ε, οικονομίας, της κινητικότητας, της ενιαίας αγοράς και επίσης για την ενότητα της αγοράς αυτή η πρωτοβουλία για την υποβολή αυτής της οδηγίας είναι άλλο ένα στάδιο πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για να καταργηθεί γιατί κυρίως καταργεί τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, των κεφαλαίων και την, ε, τα εμπόδια στη λειτουργία και την ελευθερία εγκατάστασης και επίσης λόγω των διαφορών των εθνικών ε, διαδικασιών για την ε, προληπτική αναδιάρθρωση, την αφραγκαιότητα και τη δεύτερη ευκαιρία. Και πρώτα απ' όλα είναι μια στήριξη όχι αντίθετα προσπαθεί να ενισχύσει την νομική ασφάλεια που είναι ακριβώς αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις δυσχέρειες. Αναφέρονται ορισμένες αρχές για το τι πρέπει να εφαρμοστεί με βάση την αρχή της ε, αλληλεγγύης και της ε, επικουρικότητας αλλά και με βάση την κοινή λογική γιατί η καλύτερη εφαρμογή των ε, συμφωνηθέντων των πυλώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμεθα στην εθνική και τοπική πραγματικότητα. Αυτές είναι οι αρχές της επικουρικότητας και αυτό που αποκαλώ ευφυή και λειτουργική αποκέντρωση. Αυτά όσον αφορά τις αρχές. Ο στόχος δεν είναι να παρέμβει σε αυτά που λειτουργούν σωστά, αλλά για να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο, για να υπάρχει ουσιαστική αναδιάρθρωση, να δίδεται μια πολύ σημαντική δεύτερη ευκαιρία ή αποτελεσματικές διαδικασίες σε εθνικό ή διαμεθοριακό επίπεδο. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία ασχολείται με τρία θέματα. Το πλαίσιο της προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες και τρίτον τα μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναδιάρθρωσης αφαιρεγκαιότητας και δεύτερης ευκαιρίας εισάγει σημαντικές καινοτομίε, Δηλαδή οι εταιρείε, κυρίως οι μικρομεσαίες που έχουν οικονομικές δυσχέρειες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε ότι η ΕΑΜΠΑΣ έχει πρόβλημα χρεοκοπίας. Αλλά μία επιχείρηση 50 εργαζομένων πολύ συχνά αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς ταχείας ειδοποίησης και να μπορούν να κάνουν την τάχιστη αναδιάρθρωση. Επίσης, απλοποιεί τις περίπλοκες δικαστικές διαδικασίες. Τα λεγόμενα διαδικαστικά στοιχεία κόστους που στην ε, χώρα μου αυξάνονται λόγω του κατακαιρματισμού της ενιαίας αγοράς. Θέλουμε να υπάρξει λοιπόν εξορθολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, εισάγει την ε, αναστολή των ε, ε, ιδιωτικών, των καταδεκτικών ενεργειών κατά ατόμων. Και ακόμη, υπό ορισμένες συνθήκες, όταν περάσουν τρία χρόνια, θα μπορούσε να προβλέψει και την ακύρωση χρεών για να δοθεί αυτή η περίφημη δεύτερη ευκαιρία. Η γνωμοδότηση που σας παρουσιάζουν λέει το εξής. Συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν επί της ουσίας. Αν έχω κάποια επίκριση να κάνω είναι ότι είναι ε, περιορισμένη. Θέλω να γίνουν περισσότερα για την έγκαιρη ε, προειδοποίηση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτως ώστε οι εθνικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αυτήν την ε, έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι σημαντικό να γίνεται και για την ε, αναδιάρθρωση και για την αναστολή καταδιοκτικών ενεργειών κατά του επιχειρηματία για να μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα συζήτησης ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης και ε, ζητάω να ε, δίδουν κάτι παραπάνω από μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να αποφύγουμε το κλείσιμο των επιχειρήσεων που είναι τρομερό στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να χρεοκοπήσουν οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν κάτι παραπάνω από μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ προτείνω τα κράτη-μέλη να προτείνουν στους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία με δράση στήριξης και αναγέννηση των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ασκήσουν την επιχειρηματικότητά τους. Επίσης ζητάμε η Επιτροπή να δώσει οδηγίες ούτως ώστε να υπάρχουν μια σειρά από μέτρα για να καθορίσουμε τι είναι ενέργεια ε, ανέντιμη ή κακόβουλη. Πρέπει να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα για να γίνει πιο εύκολη αυτή η διαδικασία για τα τρία που προανέφερα. Για παράδειγμα, έναντι της ε, δημόσιας δίκησης και ιδιαίτερα έναντι των ε, δικαστικών κλητήρων. Πολλές φορές αυτοί στην ουσία δρούν περισσότερο ως αρπακτικά γιατί αυτό αποφέρει περισσότερο κόστος οι, όχι μόνο οι αλλά και οι διαχειριστές των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Πρέπει λοιπόν να μετατραπούν σε κάτι που να βοηθά τις επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρχει ένας ε, δημόσιος λοιπόν κατάλογος των ε, επαγγελματιών για τους τομείς αυτούς που δεν θα πρέπει μόνο να αναφέρει κριτήρια για την ταχύτητα διάλυση μιας εταιρείας για παράδειγμα ή αλλά να αναφέρει και ποσοστά επιχειρήσεων που επανήλθαν στη βιωσιμότητα. Είναι μόνο κάποιες ιδέες. Δεν πρόκειται να αναφερθούν όλες τελικά. Η ομάδα μου αλλά και εγώ έχουμε απόψεις αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις και κατά λίγο πρόεδρε. Για παράδειγμα, ξέρω ότι πολλοί ανησυχούν για την ε, υπερχρέωση των καταναλωτών βεβαίως υπάρχουν τα αγαθά μεγάλης αξίας, για παράδειγμα ε, τα σπίτια ή τα ε, αυτοκίνητα, ιδίω αν είναι επαγγελματικά οχήματα που είναι βεβαίως χρήσιμα για την οικονομική δραστηριότητα. Αλλά αυτός ο κόσμος είναι πολύ διαφορετικός από τον επιχειρηματικό κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να κάνει τις αναγκαίες μελέτες ούτως ώστε να υπάρξει μια συγκεκριμένη οδηγία για αυτού του τύπου την υπερχρέωση. Άλλο σημείο, γιατί είναι λεπτό, είναι οι δημόσιε πιστώσει. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτύχουν την ισορροπία μεταξύ του στόχου της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης και του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος της χρηστής διαχείριση των δημοσίων πόρων. Πρέπει να δούμε τι ρόλο μπορεί να παίξει το Υπουργείο Οικονομικών για να βοηθήσει την οικονομική δραστηριότητα ή τους υπερχρεωμένους επιχειρηματίες και επίσης τα τα μη ξεπεριτούμενα δάνεια και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και καταλήγω και με συγχωρείτε που υπερεύει το χρόνο μου ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ. Τώρα. Εξ ονόματος ε, του ΕΛΚΑ, ο, ο κύριος Φαντέν Κέντελαρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως ε, υπάρχει ένα αρνητικό στίγμα περισσότερο εδώ στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ για τις εταιρείε που κλείνουν. Και βέβαια η αναγέννηση μετά από μια πτώχευση είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα όπου αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να βοηθηθούν για να στήσουν ένα νέο project. Και αυτό το σχέδιο έκθεσης θα πρέπει όντως να οδηγήσει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για την καλή πίστη. Να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας τέτοιας νοοτροπίας που να έχει στόχο την γρήγορη διάσωση αντί για την πτώχευση της εταιρεία. Αυτό είναι ένα νέο μια νέα δυνατότητα για τις χώρες, για τις επιχειρήσεις συγγνώμη, που πλέον σε βαθιά νερά και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η δυναμική ασφάλεια στην οποία βεβαιότητα στην οποία δίνει η έμφαση ο εισηγητή είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό πιστεύω πως η γνωμοδότηση που υποβλήθηκε σήμερα ακολουθεί την ε, πρόταση της Κομισιόν και γι' αυτό συμφωνούμε. Θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα για την παροχή πιο ταχείας και άμεσης βοήθειας ε, για να δίνονται ευκαιρία στους επιχειρηματίες ε, να ε, συνεχίσουν. Τώρα, όσον αφορά το κείμενο, υπάρχουν διάφορα σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να συζητηθούν και περαιτέρω και θα ήθελα να εστιάσω στο τμήμα που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους μικρούς επιχειρηματίες και τις ε, εταιρείες με ένα μόνο πρόσωπο. είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι διοικητικέ δυνατότητες για να υπάρχει δυνα... Ε, όφελος για τις ίδιες και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στους ειδικού που οφείλουν να παρέμβουν χωρίς να ε, σημαίνει αυτό άμεση νομική υποχρέωση να ξεκινήσει η διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Θα πρέπει να ανοίξει με περισσότερο η προοπτική για αναδιάρθρωση και άρα να δοθούν στα κρατημέλη τα απαραίτητα μέσα ώστε να μπορούν να προχωρήσουν. Και εδώ συμφωνώ με τα όσα είπε ο εισηγητής που μίλησε για τη σημασία ενός ε, έγκαιρου ε, συναγερμού Ίσως εδώ η Κομισιόν να διστάζει κάπως. Εμείς σας καλούμε την Κομισιόν να δρά πιο ε, γρήγορα, ταχύτερα, γιατί οι τωρινοί μηχανισμοί δεν είναι προσαρμοσμένοι στην επίλυση αυτού του προβλήματος και έτσι οι πιστωτές ή και εταιρείε να μπορούν να προστατεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Andrea Cozzolino, SD Group. Sí. Ευχαριστώ, ο Ανδρέα Κοτσολίνο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την εργασία του μέχρι τώρα. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη φιλοδοξία ορισμένων τροπολογιών που στόχο έχουν να ερμανωστούν περισσότερο οι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά σωστή διαδικασία και κοινή διαδικασία όσον αφορά το κεφάλαιο 4 και τις τροπολογίες που αφορούν καλύτερη δίκευση και εκπαίδευση των επαγγελματιών που λειτουργούν στον τομέα της αναδιάρθρωσης και της απεργιότητας. Ε, γίνονται προτάσεις για διάφορα κριτήρια και διατάξεις, ε, ώστε κάθε κράτος ε, να μπορεί να προσαρμόσει την πραγματικότητα σε σχέση με τις δραστηριότητε αυτών των επαγγελματιών. Τώρα, για τα, τις πιστώσεις, είναι απαραίτητο να προωθηθούν σημαντικά μέσα, ε, μέτρα μάλλον, όπως αυτά που προτείνονται σε αυτό το κείμενο, ας πούμε προληπτική αναδιάρθρωση, δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες ώστε να καταφέρουν να φτιάξουν μια πιο καλή διαχείριση των πιστώσεων, ήταν όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη δευτερευόντων αγορών για πιστώσεις, ώστε να αποφευχθούν οι ε, να, εγώ θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία, δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά την ανάγκη προσαρμογής αυτών των μέτρων και στα χαρακτηριστικά μάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράγμα που σημαίνει προσπάθεια για μείωση του κόστους, του διοικητικού κόστους κυρίως για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να προωθηθούν όλες οι διαδικασίες που μπορούν να εγγυηθούν τη συνέχεια, την έμεση και την άμεση τη φάση όπου μπορούν αυτά να διατηρήσουν δραστηριότητα για την επιχείρηση, τόσο όσον αφορά την διατήρηση της αξίας, προς όφελος των πιστωτών, προστασία των εργαζομένων και δεύτερο στοιχείο, ε, σχέσεις δυνάμεων σε σχέση, ε, στη διάρκεια διαδικασίας αφαιρεγγιότητας. Στο πλαίσιο της κρίσης συχνά ε, δημιουργούνται κατηγορίες και κλάσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις αρμοδιότητες για να αποφευχθεί η ε, διάλυση επιχειρήσεων. Πρέπει να προληφθούν αυτές οι καταχρήσεις, αλλά πρέπει να βελτιωθεί και το κείμενο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις ε, σχέσεις δυνάμεων, όσον αφορά την οριζόντια αναδιάρθρωση, τα μέσα ε, διαχείρισης κεφάλαιων, ώστε να αποφευθούν οι κίνδυνοι κατάχρησης και οι Θέσει υπεροχής. Πιστεύω πως είναι πολύ καλή δουλειά του εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον εισηγητή. Πολλά έχουν υποθεί ήδη, οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Σε γενικέ πολιτικές γραμμές υποστηρίζουμε τα όσα είπαν οι συνάδελφοι σκιώδεις εισηγητέ. Θα είμαι λοιπόν σύντομο και θα μπω σε λεπτομέρειες μόνο για τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι αληθεύει πως τα διάφορα καθεστώτα αναδιάρθρωσης και αφαιρεγγιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές που συνεργάζονται στην ενιαία αγορά. Άρα Θέλουμε να στηρίξουμε την ιδέα να εξετάσουμε λεπτομερέστερα αυτό το ζήτημα, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τιμωρήσουμε αυτές τις χώρες που ήδη έχουν κάνει τη δουλειά τους σωστά. Έχουν ήδη εισαγάγει καθεστώτα που λειτουργούν καλά και δεν θα πρέπει αυτές οι χώρες να τιμωρηθούν επειδή άλλες χώρες δεν έχουν αντίστοιχα συστήματα. Βλέπω όμως από το κείμενο ότι και η Κομισιόν και ο εισηγητής το κατανοούν αυτό και προτείνουν συστήματα ευέλικτα όπου είναι απαραίτητο. Δεύτερον, ήταν σχεδόν και οι τελευταίες λέξεις του εισηγητή, ε. απλώς θα τις επαναλάβω και θα τις χειροκροτήσω. Χειροκροτούμε την απόφαση του εισηγητή να μην επεκτείνει το πεδίο σε θέματα καταναλωτών, ε, υπερχρέωση καταναλωτών και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν είναι αυτός ο κατάλληλος χώρος και χρόνος. Αυτή η γνωμοδότηση δηλαδή. Τέλος, για το άρθρο 29 που αφορά στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγουν τα κράτη-μέλη για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας, θα ήταν συνετό νομίζω να δούμε ποια είναι τα πιο χρήσιμα στοιχεία και τα πιο απαραίτητα στοιχεία αλλά και ποια είναι τα στοιχεία που συλλέγονται πιο εύκολα ή πιο δύσκολα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη με επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διοίκησή τους. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Εύχομαι καλή τύχη στον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Γκουε Λόπες Περμέχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Καλβέτ Τσαμπών για την παρουσίαση και την εργασία του. Όλες οι ομάδες συμφωνούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα αφαιρεγγιότητας, ούτως ώστε μια κρίση ρευστότητας ή κάτι το περιστασιακό να μην ε, καταστρέψει μια επιχείρηση. Γι' αυτό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι είναι ένα καλό πλαίσιο για να βελτιωθεί και να απλουστευτεί η λειτουργία των διαδικασιών ε, αναδιάρθρωσης και θέτουν στο επίκεντρο την συνέχιση της ε, οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. Και άλλες επιτροπές έχουν ασχοληθεί με αυτό το σημαντικό θέμα. Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί. Πρώτον, να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, διάφορες ε, λαθροχειρίες ε, μεταξύ, για παράδειγμα, των θηγατρικών και της κύριας επιχείρησης για να θεωρηθεί ότι δεν πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ενώ είναι βιώσιμη επιχείρηση. Πρέπει επίση να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι σωστά κατά τη διαδικασία φρεγκιότητα Και τα οφειλόμενου εργαζόμενου να είναι η πρώτη προτεραιότητα και κατόπιν να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σβέν Καταρχάς να παραδεχτώ ότι στην ομάδα μας δεν έχουμε συζητήσει βάθος ε, στην ομάδα εργασίας αυτές τις προτάσεις, άρα ό,τι πω είναι τελείως ε, πρόημο. Καταρχάς χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αφαιρεγιότητα ως μέρος ε, ως τμήμα του εγχειρήματο για τις ε, κεφαλαϊκές αγορές. Αυτή η διαφορά μεταξύ των πλαισίων και ε, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αξιολόγηση του πιστοτικού κινδύνου και του πιστοληπτικού κινδύνου και έτσι ε, μειώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της αγοράς κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. παρόλο που Λοιπόν, κανείς έχει χρέη θα πρέπει να ε, μπορεί να συνεχίσει τις οικονομικές του δραστηριότητες για να μην συσσωρεύονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, σημαντικό λοιπόν είναι λοιπόν, να δούμε συγκεκριμένα στοιχεία της ε, πρότασης της Επιτροπής καλώντας για ξεκάθαρα κριτήρια σχετικά με το τι είναι η αφρέγγια δράση και η κακή πίστη ε, και πώς θα εντάσσεται κανείς στο μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς πρώιμης προειδοποίησης ε, μέσω μιας ε, κεντρικής ιστοσελίδας ενημέρωσης από την πλευρά της Κομισιόν. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς οι διαδικασίες απαλλαγής και εφαρεγγιότητας θα στηριχτούν με δεδομένα αποδείκτες που έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως ο αριθμός θέσεων που χάνονται κάθε φορά θέσεων εργασίας, επιπτώσεις στην απασχόληση και στα δημόσια οικονομικά. Παρόλο λοιπόν που η πρόταση του εισηγητή περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία, υπάρχουν τομείς που πρέπει να εξεταστούν πιο προσεκτικά. Συγκεκριμένα το κείμενο, το κείμενο περιλαμβάνει κάποιες αβεβαιότητες, δείχνει στους ε, δανειοληπτές κάποια πρόσβαση σε συστήματα πρώιμης προειδοποίησης, όμως δεν μας λέει ποια είναι αυτά τα συστήματα και πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη. Επίσης, είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα. Να εξετάσουμε πιο στενά το πώς ας πούμε θα αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι ως προς την, τα δικαιώματα ψήφου που έχουν όταν υπάρχει αναδιάρθρωση. Να μην είναι, να, είναι μια ξεχωριστή συζήτηση αυτό. Έτσι λοιπόν περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις όλων των σκιωδών και την ε, σχετική συζήτηση γιατί χρειαζόμαστε στον τομέα της ευφυαρεγγιότητας πολλούς ε, κανόνες, κοινούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδάλλως, δεν θα έχουμε την ενοποίηση των αγορών κεφαλαίου και δεν θα έχουμε τις σωστές ε, επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε το λόγο στον εισηγητή. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ζητήσει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ, παρακαλώ, εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα σας επιστρέψω το χρόνο που σας έκλεψε στην αρχή γιατί είναι αλήθεια ότι συμφωνώ με σχεδόν όλα όσα άκουσα. Όλα επικοδομητικά σχόλια, δεν βλέπω κανένα σημείο όπου να υπάρχει μεγάλη αντίφαση ε, παρά ε, διαφορετικά τα θέματα που αναφέρθηκαν συμφωνώ για όλα πρέπει να εμβαθύνουμε. Μιλάμε για ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γιατί είναι αυτές οι οποίες περισσότερο εκτίθενται στη, σε, όλα αυτά παρά οι μεγάλοι όμιλοι. Και όσα είπατε για τις αρχές επίση, ρόλος των εργαζομένων, ε, εδώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την, στην Παλώμα και στον τον εκπρόσωπο των Πρασίνων. Είμαι μέλος και της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, βλέπουμε και από εκείνη την πλευρά τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ε, θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε λοιπόν τα δύο κείμενα και ε, να υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε αυτά. Έπειτα ο Ιταλός συνάδελφος μίλησε για το δευτερόβον ε, κόστος, το κόστος και τη μείωση του κόστους για τις μικρομεσαίες και τη σχέση δυνάμεων. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε πως οι τράπεζες είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη σε όλες τις χώρες. Όμως, ε, σε πράξη είναι δυνατόν μια μεγαλύτερη συμμετοχή του δημοσίου τομέα ή άλλων δυνάμεων να μπορέσουν να, να εξισορροπήσουν και να βελτιστοποιήσουν τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας. Και γι' αυτό θα δουλέψουμε. Ο συνάδελφος μίλησε για διασυνοριακές δυνατότητες και κατά κάποιο τρόπο αυτό συμφωνεί με το όσα είπε και η κυρία Λόπες Βερμέχο Ε, όσον αφορά και τα δυσυνοριακά θέματα και την ε, FEE e, ε, λογιστική. Πρέπει να δουλέψουμε και για το benchmarking για να δούμε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργεί σωστά. Καλό είναι να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο άρθρο 29 θα το δω, δεν νομίζω ότι είναι αυτό αντιφατικό. Και στο συνάδελφο των Πρασίνων να πω ότι Πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάπως την πρόταση, πρέπει να παρακολουθήσουμε, να αξιολογήσουμε, κάπως να διευκρινίσουμε τα μέτρα, να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων που εργαζόμαστε σε αυτά σε άλλη ομάδα. Είναι μής εργασίας. Σας ζητώ όλα αυτά και όσο ακόμα ε, σκεφτείτε να τα υποβάλλετε μέσω των τροπολογιών σας για να αρχίσουμε να δουλεύουμε στις ε, συνεδριάσεις των συντονιστών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Χρονοδιάγραμμα. Έχουμε κατάθεση τροπολογιών για τις 14 Σεπτεμβρίου, εξέταση των τροπολογιών 16 Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα της Γιούρη προβλέπει την ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018. Ξέρετε ότι είναι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ και μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο και τελευταίο για σήμερα πρόγραμμα δράσης για τις χρηματοπιστικές για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εξέταση των τροπολογιών. Κύριε Λούτβικσον, εσείς ο εισηγητής και έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες υπέβαλαν τροπολογίες. Νομίζω πως αυτές εμπλουτίζουν το κείμενο. Βεβαίως ε, γίνεται η εργασία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το τελικό κείμενο θα δικατοπτρίζει τις τροπολογίες. Αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικό να φτάσουμε σε συμβιβαστική ε, ε, λύση και η Κομισιόν να ολοκληρώσει την εργασία της μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης των Κεφαλαγορών. Πρέπει επίσης η χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να ενταχθούν στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ε, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο καινοτομία και ανταγωνισμό με χρηματοπιστωτικά προϊόντα ευρύτερα που θα συμμετέχουν σε μια, σε μια εσωτερική αγορά ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων αυτών και να είναι και πιο προσιτά στον καταναλωτή. Είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη για να πάψει ο αυξανόμενος λαϊκισμός και για να βελτιώσουμε το, τις ε, προσδοκίες, μάλλον να ε, τροφοδοτήσουμε τις προσδοκίες των νέων για το ε, μέλλον. Πρέπει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση ώστε οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε να μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για του συμπολίτε μα. Έχω σημειώσει το γεγονό ότι η Κομισιόν στο πρόγραμμα δράση τη, λαμβάνει υπόψη τι προτάσει προτάσεις του, του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στο πράσινο βιβλίο για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, αλλά χρειάζεται και ένα γενικό νομικό πλαίσιο για να βελτιωθεί η διαφάνεια, να βελτιωθεί η ανάπτυξη και να μειωθούν οι φόροι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Να δούμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες μπορούν να ακυρώσουν ε, πιστωτικές κάρτες ή όταν αυτοί μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες των τραπεζών. Θα πρέπει σοβαρά να προστατεύσουμε τη νέα ζωή στο νέο κράτος μέλος για τους Ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται, πολίτες των οποίων ο αριθμός αυξάνεται. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 21ο καθεστώς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αντίθετα, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία των πολιτών με τη δημιουργία ενός πλαισίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση ας πούμε με τους ε, τραπεζικούς λογαριασμούς ή τις συντάξει. Και εδώ τονίζω τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά την μετατροπή από το ένα νόμισμα στο άλλο γιατί κάποιες φορές είναι πολύ, πολύ δαπανηρή η ε, ε, μετατροπή από το ένα νόμισμα στο άλλο και να έχουμε επίσης και μια πιο σαφή εικόνα ε, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι κοστίζει λιγότερο όσον αφορά εμβάσματα ή μετατροπές. Ακόμα ένα σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς σημαντικό στοιχείο είναι ε, ο γεωγραφικός περιορισμός. Αυτή τη στιγμή αυτό χρησιμοποιείται για να μπορέσουν ε, οι συγκεκριμένοι φορείς να διατηρήσουν κυρίαρχη θέση στην εθνική αγορά κάθε φορά. Θα πρέπει αντίθετα να μπορούν να διευκολυνθούν ε, οι δανειοδοτήσεις διασυνοριακά, ώστε ο καταναλωτής να χαίρει περισσότερο του ανταγωνισμού και να μπορεί να επιλέξει. Ε, επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη κατάρτιση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ώστε ε, ο καταναλωτής να μπορεί να προβεί ενήμερος σε, στις επιλογές τους. Τα διασυνοριακά δάνεια θα πρέπει να διευκολυνθούν με ένα κοινό ε, νομικό σύστημα όσον αφορά τέτοιου είδους πιστώσεις. Σε αυτά θα σταματήσω. Να σας πω ότι εργαστήκαμε καλά σε πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές ομάδες για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. και Όδης. Παρακαλώ. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Να υπενθυμίσω τρία σημαντικά στοιχεία για την ομάδα μου. Πρώτον, χαιρετίζουμε την ε, ρεαλιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση το σχέδιο δράση, όπως είπε και ο Σαλφος Όλε, βασίστηκε στην ε, δημόσια διαβούλευση και στην πράσινη βίβλο. Δεύτερον, δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε νομοθετήματα που μόλις ε, μεταφέρθηκαν είναι σε φάση μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία. Δηλαδή για την οδηγία για τη διανομή των ασφαλιών και την οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια. Επιπλέον θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των νέων ε, επιχειρήσεων που μπαίνουν στην αγορά και των παραδοσιακών φορέων και επιχειρήσεων που λειτουργούν. Η ομάδα μας είναι λοιπόν υπέρ των τροπολογιών που λένε ότι ο τομέας πρέπει να προσαρμοστεί στην ψηφιακή πραγματικότητα και ενθαρρύνουν το, την καινοτομία. Οι FinTech έχουν ε, φέρει επανάσταση στο χώρο. Πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε τη λειτουργία τους, όμως παράλληλα εγγυόμενοι την προστασία των καταναλωτών. Ορισμένες τροπολογίες λένε ότι πρέπει να καταρτιστούν περαιτέρω οι πολίτες. Βεβαίως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί υπερχρέωση, αλλά είναι δύσκολο. Τώρα για την ε, τυποποίηση των ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων λιανικής πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν μιλάμε για τυποποίηση. Τα προϊόντα έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες ε, της κάθε εθνικής αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε αν έχει έννοια και αν είναι δυνατόν ορισμένα προϊόντα να είναι τυποποιημένα. Η τυποποίηση ως αυτοσκοπός δεν νομίζω ότι έχει έννοια. Οι συνάδελφοι Άλντε λένε ότι πρέπει να κάνουμε μία καταγραφή όλων των εμποδίων στην εσωτερική αγορά για τα προϊόντα ε, και να κάνουμε μία σειρά από ενέργειες με το 2018. Μα το έκανε ήδη με την πράσινη βίβλο αυτό η Κομισιόν. Και η δημόσια διαβούλευση είναι αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος δράση, δράσης. Ε, αναφέρονται εμπόδια, για παράδειγμα, η τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα ή διαφορετικές κοινωνικές παροχές. Δεν έχει η Κομισιόν δυνατότητες να παρέμβει επ' αυτών. Δεν έχει αρμοδιότητα. Αυτά είναι λοιπόν τα σχόλια που ήθελα να κάνω και όπως και ο συνάδελφος Όλε αναμένω με ενδιαφέρον τις συζητήσεις με τους συναδέλφους Κιώδης. Είμαστε περίπου η ίδια ομάδα που είχε ασχοληθεί και την προηγούμενη φορά με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ashley Fox, ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τον συνάδελφο Αλέκα Μπέκ για τις παρατηρήσεις του. Η ομάδα μου έχει υποβάλει μια σειρά τροπολογίες που λένε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να βοηθάει τις καινοτόμες λύσεις, να βελτιώνει την ε, οικονομική ενημέρωση του πληθυσμού και την δημοσιοποίηση των οικονομικών πληροφοριών. Ε, δεν θέλουμε να υπάρξει μια δικτυακή πύλη της Ένωσης. Νομίζω ότι θα μπορούσε να προκαλέσει παρανοήσεις και έχουμε άλλες δικτυακές πύλες, πύλες που ήδη λειτουργούν. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες δυνατότητε, όπως μία ενιαίας επαφής για να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις λιανικής. Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υποβάλαμε τροπολογίες για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή στις οδηγίες για τις ασφάλειες αυτοκινήτων και να αντιμετωπίσουμε το θέμα ότι πολλές φορές δεν δίδονται οι αναγκαίες ε, αμοιβέ για την μη υποβολή ετοιμάτων. Δεν θα υποστηρίξουμε και ορισμένε άλλε τροπολογίε, ε, ε οδηγίε. Για να γίνουν αυτέ οι οδηγίε θα πρέπει η Επιτροπή να αποτιμήσει εάν χρειάζονται περαιτέρω οδηγίες. Η ομάδα μου θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι άλλων ομάδων για έναν ενωσιακό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Ε, δεν ε, είμαστε σίγουροι ότι χρειάζεται ένα 29ο καθεστώς για αυτά τα πράγματα. Καλωσορίζουμε την έκθεση, ευχαριστούμε τον εισηγητή και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του και με τους άλλους σκιώδης για να υπάρξουν οι αναγκαίες συμβασμοί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ινφέλτ για το Άλντε. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους που κατέθεσαν τόσο ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Όμως έλεγα και ανησυχώ, διότι παρά τις καλές προτάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως ήδη ανέφερε ο κύριος αυτή η ομάδα, όπως είπατε, εργάζεται επί αυτού του θέματος εδώ και πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι ακριβώς, δύο χρόνια ίσως. Στο μεταξύ, η τεχνολογία στις αγορές εξελίσσεται με, ταχύτατες, με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ εμείς πάμε πολύ αργά. Θα επανέλθω σε λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Κάντετ. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει καταθέσει ενδιαφέρουσε και χρήσιμες προτάσεις, αλλά δεν αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Αυτό που με απογοητεύει ιδιαίτερα και με καταθλίβει είναι ότι αυτή η συζήτηση κάθε φορά φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από το θέμα της επικορικότητας των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ για το τι θέλουμε να πετύχουμε και ιδιαίτερα με κάνει να ανησυχώ το πού πηγαίνουν οι επενδύσεις. Πάνε στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι, υπάρχουν επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ναι, αυξάνονται, αλλά είμαστε... Αλλά πόρα απέχουμε από την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι οι πιο ενδιαφέρουσε αγορές στον κόσμο. Υπάρχει ένας λόγος λοιπόν που οι επενδυτές επιλέγουν να πάνε αλλού. Αν συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση σαν μόλις να μπήκαμε στον 20ο αιώνα, θα χάσουμε και δεν εξυπηρετούμε τους πολίτες μας. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό το αιώνια θέμα της επικουρικότητας και του αν θα πρέπει να υπάρχει κάτι ευρωπαϊκό ή όχι. Ας δούμε πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε ένας κόμβος, ένα hub για τις ε, τεχνολογίες, τις χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες, τις fintech, όχι να, προ... να λέμε ότι θα κρατήσουμε την παρθενία μας όμως τελικά οι πολίτες μας να ζητούν υπηρεσίες από την Κίνα, ε, γιατί τότε πότε θα, πώς θα τους προστατέψουμε. Απάντηση στον κύριο Καντέτ. Ναι, όντως η Κομισιόν προτείνει πράγματα για να αρθούν οι φραγμοί, αλλά όχι στους βασικούς τομείς που είναι ο ε, φορολογικός τομέας, ε, η νομοθεσία κτλ. που είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην ουσία αγγίζουν μόνο περιθωριακά ζητήματα διαφάνειας, γλώσσας, τεχνικών στάνταρ που είναι σημαντικά αλλά δεν είναι η ουσία. Το πραγματικό ζήτημα λοιπόν εδώ είναι αν έχουμε το κουράγιο και τη φιλοδοξία να επιτύχουμε μια πραγματική ενιαία αγορά. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα ενιαίας αγοράς. Η ευρωπαϊκή αγορά έναντι των υπολείπων. Έχουμε λοιπόν το θάρρος και τη φιλοδοξία ή όχι. Εγώ λοιπόν, ελπίζω να έχουμε. Ευχαριστώ. Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρθηκε και δικαίως ότι ορισμένοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα των, ε, της λιανικής, ε, των λιανικών μάλλον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και είναι αλήθεια. Εγώ ε, είμαι πολύ επικριτική σε σχέση με τα όσα προτείνονται τώρα γιατί πιστεύω πως ολόκληρη συζήτηση για τις ε, λιανικές υπηρεσίες που γίνεται εδώ και τη fintech έχουν χαρακτηριστεί από μια θέση των όσων εργάζονται για τους προϋπολογισμούς και μάλλον και εργάζονται με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κέρδος παρά μόνο αν αυτό είναι εις βάρος των ε, πελατών. Μα αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποιες ήταν οι οικονομικές και οι κοινωνικές ε, συνέπειες ε, της κρίσης που ακόμα δεν έχει πάψει και αντιδρούν σε κάθε νέα καινοτομία ε, με ενθουσιασμό όπως και με ανευθυνότητα κατά τη γνώμη μου. Λέει εδώ μόνο πως ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να εποπτεύουν και να γκρίνουν αυτά τα σχέδια για να προστατεύουν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως πού υπάρχει ευθύνη, ποια είναι η ευθύνη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτές τις προτάσεις. Οι πολίτες τελικά είναι αυτοί που θα πρέπει να μετατραπούν σε ειδικού των ε, ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Και ποια είναι η απάντηση. Ε, θα έχουμε μια θηρίδα. Έχουμε ένα πόρταλ ή μια θηρίδα όπου μπορεί κανείς να αποτανθεί. Αυτή είναι τεράστια όμως ευθύνη. Έχουν υπάρξει ε, χιλιάδε καινοτομίε τέτοιε χρηματοπιστωτικέ, οι οποίε πολύ συχνά είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Άλλε τέτοιε καινοτομίε είχαν καταστροφικό αποτέλεσμα στι αποταμιεύσει ε, ε, χιλιάδων Ευρωπαίων. Οι πιο πρόσφατε συζητήσει για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα δείχνουν ότι δεν μάθαμε τίποτα από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Την προηγούμενη δεκαετία περάσαμε την κρίση λόγω της κρίσης του subprime. Τώρα γίνονται τα ίδια πράγματα μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται από το κινητά τηλέφωνα. Η προστασία των καταναλωτών δεν υπάρχει και εγώ θα συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση με την ίδια αυτή ανησυχία ώστε να αναλάβουν και τα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τις ευθύνες τους. Χρειαζόμαστε πιο συντηρητική οικονομία που να είναι υπεύθυνη και κάθε φορά που να προχωράμε, να προχωράμε ε, με, φρόνηση. Ελπίζω λοιπόν πως θα μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε πιο προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ από τους πράσινους, ο κύριος Φτασόνου. Εξ ονόματος του Γκίγκολντ που δεν μπορούσε να είναι εδώ, θα ήθελα να καλωσορίσω τις ιδέες αυτές που καλύπτονται από το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως στόχο να μειωθούν τα κόστη αλλά και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εισηγητή και περισσότερους συναδέλφους που λένε ότι αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από ε, την προσαρμογή και τον στάνταρ προστασίας ε, του καταναλωτή. Πιο φιλόδοξη δράση θα πρέπει να αναλάβει η Κομισιόν για να δημιουργήσει μια αγορά όπου οι καταναλωτέ όχι μόνο θα μπορεί να μπορούν να υποφεληθούν από τα χαμηλά κόστη, αλλά θα χαίρουν και προστασίες καταναλωτή και ποιότητα πληροφορίας ε, επί της οποίας να βασίσουν τις επιλογές τους καλύτερη οικονομία και το ευρωβαρόμετρο ε, υποτομίζουν ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά τα τέλη και τις προμήθειες ε, που μετακινούν ε, αδικαιολόγητα ποσά στις, προς τις τσέπες των, των χρηματοπιστωτικών φορέων. Και δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιε άλλε ασυμμετρίε, αλλά να ωφεληθούν οι καταναλωτέ. Έχουμε τη ιδέε τη 22, όπου καλούμε την Κομισιόν να εξετάσει όλα τους σημαντικούς φραγμούς ε, στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, ε, τροπολογία 51, υπεύθυνε επενδύσεις, καλή, έναν καλύτερο και ταχύτερη μάλλον αναφορά, ώστε να, να γίνονται ενήμερα οι επιλογές επί τη βάση ποιοτικών πληροφοριών για το βαθμό στον οποίο στηρίζουν αυτές οι επενδύσεις κοινωνικά υπεροπληκτικά project. η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών ακόμα ε, χωλένει. Έχουμε επίσης την 62 και την 121 που θα θέλαμε να λάβει υπόψη ο εισηγητής και να αναφέρω και κάποιες άλλες τοπολογίες που μπορούμε να στηρίξουμε. Με χαρά βλέπουμε ότι υπάρχει ευρεία συνένεση για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών που θα πρέπει να υπόκειται στις ανάγκες των καταναλωτών. Επίσης, καλωσορίζουμε τη στήριξη για ισότιμο πεδίο ανάμεσα στους παρόχους προϊόντων που δεν θα εμποδίζει όμως την ωφέλιμη, την, την μάλλον ρήξη 157 του κυρίου Τάγκ θα θέλαμε να συμπεριληφθεί για τα τυχερά παιχνίδια που πολλές φορές ε, είναι καμουφλαρισμένα ως ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Καλωσορίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα δράσης, αλλά καλούμε να στοχεύσει ακόμα ψηλότερα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την Μπάρμαρα Κάπελ. Ωραία. Θέλει κανείς άλλο το λόγο, όχι. Κύριε Ρούντιξον, παρακαλώ, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιτύχουμε καλές συμβαστικές τροπολογίες. Πρέπει όντως να ανταποκριθούμε στην ε, πρόκληση που είναι ενώπιόν μας. Αυτό που γίνεται τώρα με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής πρέπει να ανοίξει το δρόμο για το μέλλον. Γιατί η τεχνολογία κινείται με ραγδαίους ρυθμούς, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ε, ε αποκοπούμε εντελώς. Βεβαίως και θέλουμε αυξημένο ανταγωνισμό, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα και καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα. Και αυτό βοηθάει τους καταναλωτές αλλά πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι για το πώς ακριβώς θα επιτύχουμε αυτό μας το στόχο. Πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας ε, το συμφέρον των καταναλωτών, να έχουμε καλύτερα προϊόντα, προϊόντα που πραγματικά να βοηθούν τους καταναλωτές. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνουν τα ανοιχτά σύνορα. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να καταλήξω σε λογικές και σκόπιμες συμβαστικέ λύσεις. Φυσικά δεν στηρίζω όλα όσα προτάθηκαν, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιτύχουμε καλούς συμβιβασμούς. Ούτως ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με καλύτερο τρόπο τους καταναλωτές και τους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια στην 1η του Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Η επόμενη θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 4 ε, Σεπτεμβρίου 3 με 6.30. Ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση.